Καλημέρα σε όλες ε, και όλους. Παρακαλώ καθίστε, Οι περισσότερες είμαστε εδώ παρούσες ε, για την ψηφοφορία, έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα, καλό είναι να το σεβαστούμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές, Καλώς επανήλθατε, καλή σχολική χρονιά και εύχομαι να έχετε ξεκουραστεί. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας και ξεκινάμε με την σημερινή συνεδρίαση. Έχετε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Περνάμε τώρα σε αυτήν. Πρέπει να εγκριθεί. Υπάρχει ε, κάποια παρατήρηση επί της ημερήσιας διάταξης. Όχι. Οπότε περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Όχι. Πριν από αυτό έχω κάποιες ανακοινώσεις βλέπω. Στην συνεδρίαση της 18 Ιουλίου οι συντονιστές αποφάσισαν να συντάξουν ένα ψήφισμα και να οργανωθεί μια αποστολή στην Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για την Διευθύνη Ανάπτυξη και τον πληθυσμό 12 με 19 Νοεμβρίου 2019. Η σύνθεση της αποστολής ακόμα δεν έχει ε, αποφασιστεί. Πρέπει να λάβουμε την έγκριση στις 12 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με ένα θέμα, την παρουσίαση της δεύτερης έκθεσης για την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά της διακίνησης ανθρωπίνων όντων, όπως απαιτείται από την Οδηγία 36 2011, με τον συντονιστή καταπολέμηση τη ε, πορεία ανθρώπων. Θα σα στείλουμε εγκαίρω την ημερήσια διάταξη και επίση σα ενημερώνουμε ότι ε, υπάρχει σήμερα ένα συνεργείο το οποίο γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ και ακολουθεί την κυρία Λίσκουνκεν ε, των Πρασίνων από την Σουηδία οπότε σα ενημερώνουμε για να μην παραξενευτείτε με τι κάμερε. και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία, την ηλεκτρονική ψηφοφορία Ελπίζω λοιπόν να έχετε όλοι τις ε, κάρτες μαζί σας. Έτοιμες, έτοιμοι. Λοιπόν, βλέπετε επίσης στην ημερήσια διάταξη ότι πρέπει να γίνει η ψηφοφορία αυτή. γιατί αφορά τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το Δημοσιονομικό έτος 2020, όλα τα τμήματα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Φράνσις ε, Φιτσέραλντ και βεβαίως είναι η αρχή της νομοθετικής ε, περίοδου και θα ήθελα να πω ότι οι ψηφοφορίες για τον προπολογισμό είναι κάπως διαφορετικές από τις υπόλοιπες που πάνε τροπολογία-τροπολογία. Θα σας εξηγήσω λοιπόν τι γίνεται. Ευτυχώς ε, δεν είναι πολύ μακροσκελής. Θα αναφέρω τον αριθμό των τροπολογιών και μετά θα ψηφίζουμε. Όχι όλο τον τίτλο δηλαδή γιατί είναι σκηνοτενής και μετά θα έχετε τον αριθμό της τροπολογίας και νομίζω ότι είναι σαφές, είναι αυτεξήγητο. Ωραία. Βλέπω ότι έχουμε απαρτία. Οπότε ξεκινάει η ψηφοφορία. Τροπολογία FAM 6201. Ε, ηλεκτρονικά. Ναι, ναι. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί αφορά τον προϋπολογισμό. Οπότε θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε την 6201, την δική μας. Έχει κάποια ξεχάσει την κάρτα, έχει κάτι να πει. Όχι. Αν δεν ανάβει το λαμπάκι, ε, καθίστε αλλού, σε ένα άλλο έδρανο. Ε, εντάξει, μετά τις διακοπές μπορεί να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Α, όχι, δουλεύει. Ναι, θα περιμένω. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, θα περιμένω όμως. Ούτε εκεί έχει φως. Να, το λαμπάκι. Όχι, δουλεύει, δουλεύει. Πατήστε το κουμπί. Το πατήσατε ήδη. Α. Είναι... Είναι ακόμα αρχή της χρονιάς, πρέπει να ζεσταθούν και τα μηχανήματα. Ναι, όχι, πρέπει να πατήσετε και το δικό σας. Μόνοι σας. Ψήφισαν όλοι, ωραία, πέρας. Είμαι ε, σίγουρη ότι... Α, πού είναι ο αριθμός. Οπότε ε, είπαμε. Πρώτη μέρα μέχρι να συνηθίσουμε. Τι λέμε. Δεν γρίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Επόμενο. FAM 6202. Α, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Βλέπετε εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 6203 ΦΑΜ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενο ΦΑΜ 6204. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΘΑΜ 6205 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ΦΑΜ 6206 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ΦΑΜ 6207 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. 27 ψήφοι υπέρ. 62-08. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. 6209 και 62-10 ε, ταυτόσημες. Θα τις ψηφίσουμε από κοινό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνονται με 23 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 62-11. άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται σαφώς. Με ναι, 28 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 62-12. άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 6213, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 6214. Α, καταπίπτει. Ωραία, εντάξει. 62-15 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Φαμ. 62-18. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Μα καταπίτη ε, οι 16 και 17 εάν εγκριθεί η 15. Οπότε πάμε στην 62-18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους. 62-19. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. ΦΑΜ 6220 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται με 24 ψήφους ΦΑΜ 6221 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Με 22 ψήφους. Περνάμε στην 62-23. Άρχεται η ψηφοφορία. Καταπίπτει. Όχι, όχι. Δεν εγκρίθηκε. Οπότε παραμένει και ψηφίζουμε την 6223. Πέρας. Εγκρίνεται. Και επειδή εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει και ορίστε. Έχουμε όλες αυτές τις τροπολογίες που θα υποβάλουμε. Τελειώνει εδώ η ψηφοφορία. So, Σας ευχαριστώ. Ήμασταν πολύ πειθαρχημένοι, οπότε ε, τηρήσαμε και το χρόνο, το χρονοδιάγραμμα, πράγμα σπάνιο. Λοιπόν, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν διακριτικά, γιατί έχουμε και μια καλεσμένο, καλεσμένη εδώ, καλό θα είναι για τις εργασίες μας εδώ να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη της κυρίας Τίνα Στόλε, Γενική Διευθύντρια για τη Δικαιοσύνη και τους Καταναλωτές και να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί της ε, για τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν ε, την Επιτροπή Γυναικών να δούμε ποια είναι τα εκκρεμή λοιπόν θέματα, πού βρίσκονται οι διάφορες διαπραγματεύσεις για τους διάφορους φακέλους θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στην καλυσμένη μας, την Τίνα Στόλε και στη συνέχεια θα έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων μαζί της. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και βεβαίως από εκεί πέρα ε, οποιοδήποτε άλλος μπορεί να θέσει όποιο ερώτημα θέλει. Η κυρία Στόρα έχει το λόγο. Madam Chair, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που έρχομαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να αναφερθώ στους φακέλους που έχουν να κάνουν τις πολιτικές ισότητες των δύο φύλων στην Κοινική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Και συγχαρητήρια κυρία Πρόεδρε ε, για τη σας, τα νέα σας καθήκοντα που έχετε αναλάβει. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, όπω και στο παρελθόν με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Στο παρελθόν θα θέλαμε να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο μαζί σα, να το διατηρήσουμε, για να έχουμε μια διαστρωμένη ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να προχωρήσουν αυτοί οι σημαντικοί φάκελοι με τον οποίο εργαζόμαστε και που αφορούν ε, στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους σημαντικούς τους φακέλους που μας απασχολούν. Βία κατά των γυναικών, εξισορρόπηση επαγγελματική προσωπικής ζωής, απόκληση ε, μετα, ε, ε, ισότητα ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασία. Ε, πρώτα, η βία κατά των γυναικών όμως. Πρέπει να πω ότι το έργο για την καταπολέμηση ε, της βίας κατά των γυναικών επιγραμμικά και ε, στην πραγματική ζωή εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα της Ένωσης. Το έχετε δει και στις ε, ε προγραμματικές δηλώσεις της κυρίας Βόντερ Λάιεν. Ε, είπε ότι η στρατηγική της περιλαμβάνει ακριβώς την προτεραιότητα αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά εσείς, αλλά και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είναι πολύ στενή σύμμαχή μας σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Τα δικαιώματα των θυμάτων και η σχετική οδηγία είναι μια πολύ σημαντική νομοθετική πράξη με δεσμευτικά δικαιώματα για όλα τα θύματα βίας και βέβαια αυτό αφορά και τη βία μεταξύ των δύο φύλων. Πρόκειται για μια υπάρχουσα οδηγία που άρχισε να εφαρμόζεται ήδη το 2015, όμως τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν την έχουν εφαρμόσει πλήρως. Και η Κομισιόν χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει διαθεσή για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα την εφαρμόσουν σωστά. Δηλαδή ότι τα θύματα θα μπορέσουν όντως να ε, ασκήσουν τα δικαιώματά τους ε, όπου και να λαμβάνουν χώρα αυτή αυτά, αυτές οι εγκληματικές ενέργειες. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες παραβάση, 16 κράτη-μέλη έχουν λάβει ήδη μία ετυλογημένη γνώμη και 9 εξ αυτών έχουν φτάσει ε, στην φάση όπου έχουν λάβει μια επιστολή προεδοποιητική για να ξεκινήσει τη διαδικασία παραβάση. παραβάση. Ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν πάρει κάποια μέτρα για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους θα υποβάλουμε μια έκθεση σχετική εντός των επόμενων ημερών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των επόμενων μηνών. Αυτά σε ό,τι αφορά την οδηγία ε, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ε, στα πλαίσια μάλλον της οδηγίας των δικαιωμάτων των θυμάτων. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την παρέμβασή μας σε ό,τι αφορά την επιχραμική βία κατά των γυναικών ή την βλαπτική συμπεριφορά για τις γυναίκες. Φέτο ξεκινήσαμε ε, μια καμπάνια στα media, ένα hashtag respect for her, σεβασμός για αυτήν, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στη δημόσια ζωή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο που ε, φιλοξένησε την ε, αφετηρία αυτής της καμπάνιας και τη σχετική εκδήλωση. Έχουμε ξεκινήσει ε, επαφές και με πλατφόρμες κοινωνικών ε, μέσων δικτύωσης. Ε, Υπάρχει ένας κώδικος συμπεριφοράς ε, για την παράνομη, τον παράνομο λόγο μίσου επιγραμμικά από το 2016 και τώρα που εργαζόμαστε επί αυτού του θέματος ε, της επιγραμμικής βίας ε, αυτό το ο κώδικα συμπεριφορά είναι το μοντέλο για μας συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, συμμετέχει και ο καθημαϊκός κόσμος στην προσπάθεια αυτή. Έως τώρα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την επιγραμμική βία των γυναικών, όμως υπάρχουν κάποια σημεία σε διάφορες ε, νομοθεσίες σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και σε επίπεδο κρατών που ε, καλύπτουν το θέμα αυτό. Η σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολη μια πολύ σημαντική σύμβαση στον τομέα αυτών, απαιτεί από όλα τα συμβαλόμενα μέρη να ποινικοποιήσουν ε, την βία κάτω γενικών επιγραμμικά και όχι μόνο, ε, καθώς και την ποινικοποίηση της ε, παρενόχλησης. Και έχουν πολλά τα μέλη αυτής της σύμβασης. Αυτές οι χώρες έχουν ήδη ποινικοποίησει πολλές μορφές βίας κατά των γυναικών. Βεβαίως ποικίλει η εφαρμογή από τη μία χώρα στην άλλη. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι νομικές διατάξεις που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Και εδώ προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και την ελευθερία ε, έκφρασης βέβαια. Θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε το έργο αυτό ε, αντιμετώπισης της γραμμικής ε, βίας κατά γυναικών με άλλες εργασίες που έχουν να κάνουν με, την, με το παράνομο και βλαβερό ε, περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης χρειαζόμαστε καλύτερα στατιστικά στοιχεία αυτό είναι πάντα η βάση των εργασιών μας. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ισχύει. Η Eurostat έχει αρχίσει να... μια έρευνα το 2016. Έγινε πρώτα μια πιλωτική το 2008-2019 σε κάποιες χώρες, 12 χώρες. Θα γίνει και μια πλήρης έρευνα του χρόνου. Το Σεπτέμβριο του 2022 θα έχουμε τα αποτέλεσματα το αργότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξορρόπηση επαγγελματική και προσωπική ζωή. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γυναικών, ε, την Επιτροπή ΦΑΜ για το έργο της από κοινού ε, με εμά έτσι ώστε να περάσει η συγκεκριμένη οδηγία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ε, ένα κομβικό σημείο, εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου και προβλέπει μέτρα έτσι ώστε να μοιράζονται τα καθήκοντα στο σπίτι ε, για να μπορούν και οι γυναίκες ε, να συμμετέχουν πιο ισότιμα στην αγορά εργασίας. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη θα είναι υπεύθυνη για να βοηθήσει τα κρατημέλη να εφαρμόσουν του κανόνε αυτού. Θα λάβουν χώρα εργαστήρια για να του καθοδηγήσουμε και θα έχουμε και μια συνεδρίαση εναρκτήρια για τι εργασίε αυτέ πριν από το τέλο του έτου. Οι εργασίε αυτέ χρειάζονται και χρήματα. Υπάρχει και το πρόγραμμα για την ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ των πολιτών και εκεί περιλαμβάνεται το θέμα της ε, επαγγελματική και προσωπική ζωής. Ε, θέλουμε να καταπολύσουμε τα στερεότυπα. Θέλουμε επίσης πολιτικές που να είναι φιλικές προς τις οικογένειες εντός των επιχειρήσεων. Θα ενισχύσουμε την εφαρμογή ε, των εκστρατιών, των καμπάνιων ε, και θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα νέα τους δικαιώματα όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή των σχετικών νομοθετημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα. Ε, είναι η βάση πολλών εκ των δραστηριοτήτων μας αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα το οποίο χρονίζει είναι η διαφορά η μισθολογική. Μειώνεται βέβαια αλλά πάρα πάρα πολύ αργά και ζητήθηκε από την Κομισιόν να πάρει μια νομοθετική πρωτοβουλία για ζητήματα διαφάνειας μισθολογικής. Ξέρετε ότι η αρχή σύμφωνα με την οποία οι άντρες και οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν την, τον ίδιο μισθό, τις ίδιες απολαβές για την ίδια εργασία ή για εργασία ίδιας αξίας υπάρχει από το 1957 στη συνθήκη. Μετά από 60 χρόνια όμως αυτό το χάσμα το μισθολογικό είναι 16% Δηλαδή οι γυναίκε λαμβάνουν 16% λιγότερο από του άνδρε. Ε, και αυτό που είναι ακόμα πιο ενισχυτικό είναι ότι η, η απόκληση σε ό,τι αφορά τι συντάξει είναι στο 35%. Και αυτό δείχνει την χρόνια ανισότητα, την ανισότητα μια ζωή, αν θέλετε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διότι οι γυναίκε αναγκάζονται να σταματήσουν την καριέρα του συχνά κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία για να καλυφθεί αυτό το χάσμα και το πρώτο βήμα θα είναι ένα βήμα που αφορά στη διαφάνεια. Ε, με, τις δράσεις, με τη δράση διαφάνειας ε, θα γίνει πιο ορατή ε, αυτή η διάκριση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε από τους εργοδότες να μας δώσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία ανάλογα με το φύλλο. Ήδη στον Ηνωμένο Βασίλειο είδαμε ότι η σχετική νομοθεσία περί νομοθεσίας τη μισθολογικής ε, ανέδειξε εντυπωσιακέ διαφορές μισθοδοσία σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως το BBC παραδείγματο χάρη. Η διαφορά στα μπόνους επίσης ήταν τη τάξη του 60-70% σε κάποιες ε, εταιρείε ε, μεταξύ των δύο φύλων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνει η χώρα μια αξιολόγηση των νέων κανόνων και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η νέα επικεφάλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δεσμευτεί στα πρώτα 100 στις πρώτες 100 μέρες της θητείας της να προετοιμάσει μια νομοθεσία για την ε, μισθολογική ισότητα ξέρουμε, και τη, μάλλον για τη διαφάνεια ε, σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία, αλλά αυτό βέβαια δεν αρκεί. Το γνωρίζουμε. Ε, θα πρέπει να το δούμε ευρύτερα το θέμα, ε, να δούμε ε, άλλες μορφές διακρίσεων που υπάρχει σε χαμηλότερε ε, χαμηλότερες μισθολογικές κατηγορίες. Τώρα για το gender mainstreaming. Θα ήθελα να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργαζόμαστε στο ζήτημα αυτό διτά έχουμε συγκεκριμένε δραστηριότητε, συγκεκριμένε δράσει, αλλά εφαρμόζουμε και το gender mainstreaming, έχουμε υπάρχει μια task force στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου συμμετέχουν σχεδόν όλε οι γενικέ διευθύνσεις και θέλουμε ε, αυτή την ατζέντα να την προωθήσουμε σε όλου του τομεί ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ζήτημα που εδώ και καιρό είναι επιτάπητο είναι οι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια. Είναι ένα θέμα το οποίο εδώ και πολύ καιρό είναι έχει κάπως κολλήσει. Η πρόεδρος είπε ότι στι πολιτικέ κρατικέ γραμμέ τη θα προσπαθήσει να βρει μια πλειοψηφία για να μπορέσει να απεμπλακεί η συγκεκριμένη οδηγία και εδώ υπάρχει υποστήριξη από το Κοινοβούλιο. Χωρίς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε κάποιες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο αλλά αυτές οι εξελίξεις προχωρούν με άνισο τρόπο. Ευρωπαϊκή νομοθεσία λοιπόν θα ήταν κάτι θετικό εδώ και βεβαίω θα συνεργαστούμε στενά και μαζί σας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα τελειώνοντας θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη στρατηγική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ξεκινήσαμε την προπαρασκευή της στρατηγικής αυτής. Ταυτόχρονα αξιολογούμε τις στρατηγικές δεσμεύσεις και τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας ε, προσπαθούμε λοιπόν να βασιστούμε να οικοδομήσουμε πάνω στα διδάγματα της προηγούμενης περίοδου θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα απαντήσουμε στα ζητήματα τα νέα που προκύπτουν και τις ε, εξελίξεις. Έγινε να χώρα μια δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσουμε το έργο που έχει λάβει η χώρα στα πλαίσια των στρατηγικών δεσμεύσεων. Ε, από 8 Μαρτίου ως τέλος Μαΐου έλαβε χώρα αυτή η δημόσια διαβούλευση και θα δημοσιεύσουμε σύντομα τη σχετική έκθεση. Η Επίτροπος Γιούροβα έχει στείλει και μια επιστολή στους συναδέλφους της ρωτώντας τους τι έχουν κάνει για να πετύχουν μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των δύο φίλων στις δικούς τους τομείς δραστηριότητα και τι θεωρούν ότι ακόμα μένει να γίνει και βεβαίω οι δικέ του απαντήσει ε, θα τροφοδοτήσουν τι εργασίε μα. Υπάρχει και μια συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα των δύο φύλων. Συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, η κοινωνία των πολιτών, οι κοινωνικοί εταίροι και η δική του συνεισφορά επίση θα μα βοηθήσει. Υπάρχει και ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων για ζητήματα ισότητα μεταξύ των δύο φύλων που επίση αξιολογούν του διάφορου αυτού τομεί. Και ένα εμπειρογνώμονα από αυτό το δίκτυο προετοιμάζει μια εκτίμηση τη στρατηγική δέσμευση η οποία θα είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο λογικά. Ε, έχουμε λοιπόν πολύ υλικό και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη στρατηγική 2020 με βάση το υλικό αυτό ε, που θα καλύπτει μεταξύ άλλων και θέματα τα οποία αναφέρθηκαν και στις πολιτικές κρατικές γραμμές βία των γυναικών, ε, διαφάνεια στην απασχόληση, ε, συμμετοχή των γυναικών στα ειδικά συμβούλια, ισορροπία μεταξύ οικογενειακή και επαγγελματική ζωής κτλ. Έχουμε μια στρατηγική λοιπόν φιλόδοξη που θα μα βοηθήσει να προχωρήσουμε γρήγορα ε, προς μεγαλύτερη ισότητα των δύο φύλων. Αυτά από μένα είμαι έτοιμη για να απαντήσω στα ερωτήματά σα ελπίζω. Uh, Uh, your... Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευρύτατη αυτή επισκόπηση Όπω είπα, θα δώσω το λόγο σε όλου του συναδέλφου που ενδιαφέρονται, ξεκινώντα από του συντονιστέ. Μετά θα ακούσουμε του υπόλοιπου συναδέλφου και μετά τι απαντήσει τη κυρία Αστόλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σα και τη δουλειά που κάνατε. Καθώ και τη συνεργασία σα με την Επιτροπή μα. Είναι τόσο πολλοί τομεί που αναπτύξατε και μπαίνω σε πειρασμό να του δείξω όλου, αλλά θέλω να σταθώ σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία. Για τη βία κατά των γυναικών. Σίγουρα εδώ δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δείξουμε επίκαια. Έχουν υπάρξει αλλαγέ ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια στην ε, παιδεία, αλλά δύο ζητήματα αναδεικνύονται σημαντικά. Από νομοθετική σκοπιά, τι μπορούμε να κάνουμε για τον έλεγχο. Γιατί υπάρχουν θέματα βίας όπως οι γενεκοκτονίες που είναι πολύ σοβαρά όσο προς την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Ε, πολύ ωραίο να έχουμε οδηγία, όμως θέλουμε και στην πράξη να δούμε πώς εφαρμόζεται. Χρειάζεται πάρα πολύ κατάρτιση. Χρειάζεται οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς να εκπαιδευτούν, η αστυνομία, τα δικαστήρια. Οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί πρέπει να αλλάξουν οτροπία. Είναι πολύ λοιπόν η δουλειά που χρειάζεται. Και μας ενδιαφέρει τι να αναλαμβάνετε για να το υποστηρίξετε αυτό. Για το μισθολογικό χάσμα. Ως προς το, τη μισθολογική αυτή απόκληση. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ τη δουλειά που κάνατε για την διόρθωση του προβλήματος αυτού. Είπατε ότι είναι ε, ε, κρίσιμη σημασία ε, οι ίσε αμοιβέ. Και ότι κυρίω πρέπει να υπάρξει νομοθεσία για την καταγραφή των στοιχείων περί απόκληση. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν. Συμφωνώ. Και εν τέλει να πω ότι εύχομαι η υπηρεσία σας να υποστηρίξει κοινέ πρωτοβουλίε με την δική μα την Επιτροπή και άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, διότι πολλά από αυτά που κάνουμε πρέπει να είναι διατομεακά. Όχι μόνο στο επίπεδο που λειτουργούμε εντό τη Επιτροπή αυτή, αλλά και σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων. Πρέπει να δούμε πρωτοβουλίε που να έρχονται από. Ε, που να υποστηρίζουν τα δίκαια των γυναικών, ε, που να έρχονται από εσά και από άλλε γενικέ διευθύνσει ή κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να γίνει και αυτό. Ε, Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα θα ακούσουμε κάμποσε ερωτήσει και μετά τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα σχόλια, ευχαριστώ και για την δουλειά σας. Είναι θαυμάσιο το ότι μια στιγμή... Ε, δεν με ακούτε? Λοιπόν, Είναι βεβαίως πάρα πολύ καλό το ότι εσείς από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης αναζητείτε επαφή με τις άλλες ε, επιτροπές. Γι' αυτό ακριβώς ε, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες και άνδρες που λένε ναι εντάξει καλά είναι αυτά αλλά λίγα. Και βεβαίως είναι στο DNA μας να μην είμαστε ικανοποιημένοι εδώ μέσα, αλλά να συνεχίσουμε. Αλλά θα ήθελα να σας επενέσω. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε κάτι το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, είναι το θέμα των κυρώσεων. Έχουμε το θέμα γυναίκες στα δουσού, το θέμα του μισθολογικού χάσματος, ε, την πρόληψη της ε, βίας, ε, αλλά και το τι γίνεται όταν ασκηθεί βία. Γιατί οι κυρώσεις είναι τόσο περιορισμένες. Θεωρούν, ε, νομίζω οι άνθρωποι, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι κυρώσεις. Ε, δεν κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό. Ε, για να δούμε τι θα γίνει και με την εφαρμογή της συνθήκης Κωνσταντινούπολης και ε, δεν εννοώ να, να επιβάλλουμε κυρώσεις στις χώρες, ε, αλλά να υπάρξει κάποια ποινή των δραστών. Νομίζω είναι θέμα και του κοινού περί δικαίου αισθήματο. Αλλιώ θεωρείται ο τομέα αυτό κάπω πιο ήπιο. Και θα ήθελα να πω κάτι ω ε, Γερμανίδα. Εγώ ντρέπομαι για το ότι η Γερμανίδα η Γερμανία εφάρμοσε τη σχετική οδηγία ε, για τι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια στο εσωτερικό, αλλά το μπλοκάρει στην Ευρώπη. Ε, δεν γίνεται και ντρέπομαι ως ε, Γερμανίδα βουλευτής. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να συμβαίνει και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείτε τι συμβαίνει στην κάθε χώρα αφενός και πώς ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί πέρα προκύπτει ότι υπάρχει μια στρατηγική σε συγκεκριμένα σημεία να καταψηφίζουν πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το ότι τα εφαρμόζουν στο εσωτερικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οδηγία αυτή. Η, Γερμανία το εφάρμοσε κατόπιν της ε, συμφωνίας των κυβερνητικών εταίρων αλλά το μπλοκάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και για να τελειώνω τώρα χρειαζόμαστε ξανά μια στρατηγική, στρατηγική ισότητας και δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή παρακαλούσαμε την προηγούμενη φορά, 25 υπουργοί το ζητούσαν να υπάρξει μια στρατηγική και δεν υπάρχει. Έχουμε ένα κενό 5 ετών στην παρακολούθηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακολουθήσω να σας παρακαλέσουμε συγχωρείτε, να κάνετε ό,τι μπορείτε εντό των δυνατοτήτων σας για να αποκτήσουμε μια στρατηγική ισότητα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Δίνω τον ε, λόγο τώρα στην ε, συναλφό του Ρινιού. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε που ήρθατε. Συμφωνούμε με όσα είπατε. ιδίω για τα σημεία που αναφέρατε, τη βία των γυναικών, την ε, μισθολογική απόκληση και την εξισορρόπηση επαγγελματικού και γενιακού βίου. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες νομοθετικές πράξεις σε αρκετές χώρες, όμως αυτό που λείπει είναι η δράση σε κοινοτικό επίπεδο. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε ως ιδέα είναι ένα είδος συμφώνου Σιμών Βέγη. Δηλαδή να καταγράψουμε τι νομοθετικές πράξεις υπάρχουν στις διάφορες χώρες ήδη και να κοιτάξουμε η ισχύ του να επεκταθεί σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να μην χρειαστεί να επινοήσουμε κάτι όταν κάποια πράγματα ήδη λειτουργούν καλά. Και ακριβώς επειδή κάποια πράγματα λειτουργούν καλά, αυτό που μας λείπει ενδεχομένως είναι δείκτες, δείκτες ε, αριθμητικοί. Σήμερα, εάν θέλουμε να δούμε με τις διάφορες οδηγίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι συμβαίνει, αυτές που υποτίθεται ότι καθορίζουν την μισθολογική ισότητα. Υπάρχουν ε, μελέτες αξιολόγησης. Υποτίθεται ότι μπορούμε να δούμε πώς προχωράει η κατάσταση και πού έχουμε κάνει πρόοδο. Ας το δούμε λοιπόν. Για να είναι ακριβείς και ορθολογικές οι πληροφορίες μας. Είναι καλό ε, να μπορεί κανείς να, να, μπορεί να υποστηρίξει όλα αυτά με αριθμούς. Και μετά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών. Σήμερα μας μιλήσατε για τις δικές σας τις αρμοδιότητες, το δικό σας το τομέα. Όμως αυτό ο τομέας έρχεται και αρχίζει να λειτουργεί μετά την εφαρμογή άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Ένα παράδειγμα, το εράσμο. Το Εράσμους αφορά Ευρωπαίους φοιτητές που θέλουν να έχουν μια καλύτερη επαγγελματική προοπτική από αυτούς που δεν ε, πήραν ποτέ μια υποτροφία εράσμου. Στο Εράσμους ας πούμε υπάρχει ισότητα γυναικών ανδρών, το παρακολουθούμε, υπάρχουν στοιχεία. Πού είναι η συνοχή λοιπόν σε σχέση με την εφαρμογή των διάφορων ευρωπαϊκών πολιτικών μέχρι να φτάσουμε στα στοιχεία που τελικά αφορούν τη δική σα γενική διεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Κόνκε νομίζω δεν είναι εδώ. Με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα μεταξύ των γλωσσών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα από την κυρία, από ε, την, κυρία Άντερσεν. Δεν βλέπω να είναι εδώ. Η κυρία Βυσνιεύσκα. Δεν νομίζω ότι είναι στην αίθουσα, η κυρία Σάντρα Περέρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις. Η οικονομική κρίση έπληξε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που έφερε φαινόμενα φτώχειας, ε, κοινωνικής ανισότητας και ιδίως στι γυναίκες της περιοχής της Υπέθρου η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θέλει να, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη φτώχεια και αυτές τις μισθολογικές αποκλήσεις και τις διαφορές μεταξύ των φύλων. Δεύτερη ερώτηση. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει μια σαφή τοποθέτηση ως προς την σεξουαλική εκμετάλλευση και την ε, ε, εκπόρνευση. Ε, θα συνεχίσετε να συνεργάζεστε, να συνεργάζεστε μαζί μας για να καταπολεμήσουμε την επόρνευση, την πορνογραφία και την βία κατά των ενήλικων γυναικών και κοριτσιών. Το Κοινοβούλιο έχει μια σαφή τοποθέτηση για την υγεία και τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την θέση των γυναικών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιτρέψουμε νόμιμες και ασφαλείς ε, διακοπές κοίησης, αμβλώσεις και οι γυναίκες να μπορούν να κάνουν το δικό τους οικογενειακό και ένα παραγωγικό σχεδιασμό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αστόλα θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας τώρα και μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πολύ. Και με αυτές τις ερωτήσεις και μόνο βλέπουμε πόσο ευρύ είναι το πεδίο που καλύπτει η συζήτησή μας και πόσο περίπλοκο. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την Επιτροπή στο σύνολό της, όπως προείπα. Πρώτα απ' όλα για τον υποχρεωτικό έλεγχο. Κάτι που το ανέφερα και στην αρχή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα για τα φύλλα. Εκεί, για κάποιο λόγο, είναι που φωλιάζει η αρχή της βίας, των φαινομένων βίας. Για την επιγραμμική βία κατά των γυναικών. Αυτό φοβίζει, τρομάζει γενικώ τον ε, κόσμο και μιλάμε για απλούς πολίτες που δεν θέλουν να κάνουν πολιτική καριέρα, θέλουν όμως να έχουν την ελευθερία της έκφρασής τους στα κοινωνικά δίκτυα. Και μετά δέχονται επιθέσεις και τους παρενοχλούν. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ως προς τα θύματα και την εκπαίδευση φορέων, υπηρεσιών, υπαλλήλων και με κυβερνητικών οργανώσεων. Πολλά από αυτά ήδη γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Μπορούμε κι εμείς κάτι να κάνουμε με τα κονδύλια που διαθέτουμε στη γενική μας διεύθυνση. Μπορούμε να ενισχύσουμε για τις κοινέ πρωτοβουλίες. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι δεν είναι τα πάντα θέμα νομοθεσίας. Πολλοί από αυτή τη δουλειά είναι θέμα άλλων δράσεων, κοινέ πρωτοβουλίε, κοινέ εκδηλώσει, νομίζω ότι ήδη είχαμε και φυσικά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σα. Κυρώσει. Δύσκολη ερώτηση. Τα κράτη-μέλη έχουν δικά τους ποινικά συστήματα, διαφορετικά βασίζονται σε διαφορετική δομή και διάρθρωση. Το επίπεδο των κυρώσεων από κάτω μέλο σε κράτο μέλο είναι διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλες οι κυρώσει πρέπει να είναι ακριβώ οι ίδιε εξορισμού. Πρέπει να προβλέπονται στο σύστημα σε ένα κατάλληλο, ορθό επίπεδο. Αυτό μα ενδιαφέρει και κοιτάμε να ελέγχουμε. Τώρα να τονίσω την ανάγκη να ενισχύσουμε τη διάσταση της πρόληψης. Όταν μιλάμε για γυναίκες, μιλάμε για έμφυλη βία, βία κατά των γυναικών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τους άνδρες. Καταπολέμηση στερεοτύπων είναι το θέμα πάλι. Πώς θα βοηθήσουμε τους άνδρες να καταλάβουν περισσότερα. Μερικοί ξέρω ότι μετά τι πράξει βία αισθάνονται χάλια και δεν θέλουν να συνεχίσουν, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν. Πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε για τις γυναίκες στα συμβούλια των επιχειρήσεων. Ε, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε με αυτό και έχει γίνει ήδη κάποια πρόοδος. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σε επίπεδο κρατών μελών. Οι προτάσεις ήδη είναι επιτάπητος. Ήδη κάτι έχει γίνει και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ακριβώς με τη δήλωση ότι η δουλειά παρεκολύθη κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού. Ξέρω ότι εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της περασμένης θητείας και υπήρξε στι ε, στις προθέσεις σας ανάγκη μεγαλύτερης προβολής από αυτή που τελικά έχει η στρατηγική μας. Χαίρομαι πολύ που η πρόεδρος της Επιτροπής τώρα είπε ότι θα ε, γίνει πράξη η στρατηγική στατιστικές και βέλτιστες πρακτικές. Είναι η αρμοδιότητα της ΕΙΓΕ, του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, με τους οποίους θα συζητήσετε και αργότερα, να προσφέρουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία με δείκτες για τον τομέα αυτό και νομίζω ότι έχουμε πολύ υλικό στα χέρια μας. Είναι εν μέρη θέμα και μέρος της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Κάποιοι απλώ δεν τα γνωρίζουν. Ακόμη και για το μισθολογικό χάσμα και το συνταξιδοτικό χάσμα. Το 35% είναι ποσοστό που σοκάρει. Όταν ε, η πληροφορία αυτή, ο αριθμός αρχίζει να διαδίδεται, να γίνεται γνωστός, τότε ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί οι στατιστικές, λόγου χάρη, στα προγράμματα Εράσμους και το πώς ε, κατανέμονται τα ποσοστά μεταξύ νεαρών ανδρών και γυναικών, δεν ξέρω αν υπάρχουν στατιστικές για τα αγόρια και τα κορίτσια στο Εράσμους. Δεν μπορώ να σα το επισκεφθώ. Δεν μπορώ να σα το υποσχεθώ. Άλλες στατιστικές μου φαίνονται σημαντικότερες. Έχουμε και άλλες για το τι κάνουν οι νέοι σε διάφορους τομείς. Υγεία των γυναικών, αναπαραγωγικά δικαιώματα. Ένα πράγμα πρέπει να τονίσω εδώ. Η νομοθεσία περί οικογενειών, το οικογενειακό δίκαιο, συνεχίζει να είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Ε, άπτεται της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Το ζήτημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο που πηγαίνει από ένα σημείο σε κάποιο άλλο. Πώς θα μπορέσει να διατηρήσει τα δικαιώματά του ο κόσμος αυτός. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κοκκινάκο δίκαιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά μπορούμε να κάνουμε από το επίπεδο του τομέα της δικαιοσύνης. Ελπίζω να απήντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ και να συνεχίσουμε. Θα διαβάσω τώρα απλώς τα ονόματα, τον κατάλογο των αγορητών Δεν νομίζω θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μα, αν όλοι μιλήσουν πολύ. Αλλά επειδή είναι η πρώτη μα συνεδρίαση στην Επιτροπή μετά το καλοκαίρι, καλό είναι να ακολουθήσουμε το παχκούχ των θεμάτων που βρίσκεται επιτάπητο και να τα δούμε εκτενώ. Διαβάζω τα ονόματα. Μίλα, Μέλχιο, Τζόουν, Λιτάου, Μαρκέ, ε, ε, Πλίνκεβιτσούτε, Παλόπ, Γκάλβε Μουνιό, Ελέν Φρεζόν, Βλέπετε ότι είναι πολλοί αυτοί που θέλουν από εμά να θέσουν ερωτήσεις. Οπότε η έκκλησή μου είναι παρακαλώ σύντομα. Κάπως πρέπει να κλείσουμε το θέμα. Ο λόγος στη Ραφαέλα. Yes. Α? Yes, thank you very much. Yes, it was a surprise for me too that I... Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, και εμένα προξένησε έκπληξη ότι είμαι η πρώτη. Το ερώτημά μου είναι το εξή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σα Και χαίρομαι που αναφερθήκατε στο θέμα των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και από όταν έγινα σκιώδη συγγήτρια ε, με απασχολεί το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι συγκεκριμένα θα κάνει η Κομισιόν για να ξεμπλοκάρει το ζήτημα αυτό. Στατιστικά στοιχεία από την Ολλανδία χτες δείχνουν ότι το ποσοστό των γυναικών στα ΔΣ μεγάλων εταιριών έχει ανέβει αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλό και όχι μόνο στην Ολλανδία και νομίζω έχει φτάσει η στιγμή ναι, να προχωρήσει το θέμα, αλλά θα ήθελα να μάθω τι συγκεκριμένα θα κάνετε για να ξεμπλοκάρει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, τι θα κάνει η Κομισιόν για να προωθήσει αυτό το θέμα. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο εν τω μεταξύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Τζάκι Jones. Α, συγγνώμη. Κυρία Μελχιόρ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Αναφέρατε την βία κατά των γυναικών. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο ερώτημα της κυρίας Fitzgerald για τον καταναγκασμό και την ψυχολογική βία. Γιατί η σωματική βία κατά των γυναικών ε, και η ενδοοικογενειακή ε, συχνά, συχνότερα είναι ε, άνδρες ε, κατά γυναικών ε, αλλά συνήθως έχει προηγηθεί ψυχολογική βία και πίεση. Τι θα γίνει λοιπόν. Κάποια κράτη-μέλη το έχουν ποινικοποιήσει αλλά υπάρχει δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα. Επίσης για το ίδιο θέμα ένας κοινό παρονομαστής μεταξύ τρομοκρατών και λοιπόν είναι ότι έχουν ασκήσει βία σε γυναίκες στο περιβάλλον τους. Τι κάνει η Κομισιόν σχετικά και επίσης ε, θα ήθελα κάποια καλύτερα στατιστικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φαίνονται οι γυναίκες ε, κάπου στα στοιχεία αυτά. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομοι. Τζάκι Jones, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Τέσσερα θέματα έχω, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε φέτος 25 χρόνια από την πλατφόρμα του Πεκίνου και επίσης ε, την 40η επέτειο του Σίντολ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν κάνει κάτι η Κομισιόν ε, με βάση την νομοθεσία αυτή. Παράδειγμα του χάρη. Έχουμε μια ευρύτατη σύμβαση, αγγίζει όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέραμε ήδη, αλλά κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως είναι ακριβώς το να το εντάξουμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Παραδείγματο χάρη μας επιτρέπει ε, η σύμβαση ΣΥΝΤΟ να δούμε, να φέρουμε και στο εσωτερικό κάποια μέτρα τα οποία θα επανορθώνουν και τις αδικίες του παρελθόντος. Ε, παραδείγματος χάρη ε, την ανισότητα στο αποτέλεσμα, αυτό το οποίο αναφέρατε για τις ε, συντάξεις παραδείγματος χάρη οι παλαιότεροι νόμοι σημαίνουν ότι οι γυναίκες έχουν σήμερα χαμηλότερες ε, συντάξεις αν δείτε υπάρχει και μια υπόθεση που εκκρεμεί στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούμε λοιπόν να έχουμε εδώ πέρα μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων που θα βασίζεται σε κάποιες τέτοιες αρχές αυτά τα δύο μετά Χαίρομαι για αυτό το οποίο είπατε για τις γυναίκες ε, στα ΔΣ. Ξέρετε ότι οι Ευρωπαίες δικηγόροι ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Έχουμε πάει σε 180 γενικές συνελεύσεις ανωνύμων εταιριών ε, ακριβώ ε, για να θέσουμε αυτό το ζήτημα. Επίσης χάρηκα που χρησιμοποιήσατε ένα παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά τις δύσκολες αυτές ώρες η διαφάνεια λοιπόν λειτουργεί, αλλά θα ήθελα να σκεφτείτε και το τι γίνεται μετά. Γιατί η διαφάνεια αυτή πρέπει να είναι πλήρης ε, και να υπάρχουν και συνέπειες για το ότι δεν υπάρχει είτε διαφάνεια είτε υπάρχει, ε, υπάρχουν άνεσες αμοιβέ. Και τέλος, θα ήθελα να σας παρακαλώ να δείτε το θέμα της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, ειδικά των κοριτσιών που υφίστανται τις περισσότερες ε, διακρίσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαγγέλ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την προσέλευση της κυρίας Αστόλα για να μας παρουσιάσει την πολιτική της Επιτροπής για αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική. Μια ερώτηση απλώς και μια παράκληση για την διατήρηση της ισορροπίας επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, ένα από τα σημεία που αναδείξατε ανάγλυφα στην παρουσίασή σας. Εξαιρετική εμπειρία είχαμε για τη δημιουργία αυτού του προτύπου της προδιαγραφής που θα πρέπει να διέπει τη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων και να συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό. Έχουμε 58 φορείς που ασχολούνται και εφαρμόζουν το πρότυπο αυτό και έχουν πιστοποιηθεί οι περισσότεροι. Είναι πολύ σημαντικό ε, το πρότυπο αυτό, η προδιαγραφή αυτή, διότι το αντίθετο στην πράξη πραγματικά διαταράσσει την ισορροπία μιας επιχειρήσης. Μιας Ήθελα λοιπόν να κάνω την εξή ερώτηση. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια διαδικασία ευρωπαϊκής προδιαγραφής για την διατήρηση της ισορροπίας οικογενειακού επαγγελματικού βίου. So, thank you very much. Uh, Eugenia, uh... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορτίδα, α, συγγνώμη. Ε, όλο μπερδεύω τη σειρά. Όμως τώρα θα μιλήσει πρώτα η κυρία Μπλενκεβιτζιούτα. Ε, εσείς ετοιμαστείτε εντωμεταξύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Θέλω να διαβάσετε τις ευχαριστίες μας προς όλους τους συνεργάτες σας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οδηγία, μιας και η πρωτοβουλία σχετικά με την οδηγία αυτή προέρχεται από τη δική μας Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αυτό το σχέδιο οδηγίας η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν βεβαίως πολύ πιο φιλόδοξη και σας ζητώ να συμπεριλάβετε να κάνετε ό,τι μπορείτε ε, στην προσπάθειά σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορούμε να απαιτήσουμε πραγματικά να μπορεί να αποζημιώνονται, να υπάρχει μια πληρωμή για τα εξαρτώμενα άτομα και την περίθαλψή τους από γυναίκες. Αγιώς δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση για τις γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Σας ζητώ λοιπόν να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση ε, στους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν, να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία έτσι ώστε να λάβουν χώρα πραγματικές αλλαγές. Χαιρετίζω την δέσμευση που ανέλαβε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση ε, του μισθολογικού χάσματος εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της. Βεβαίως δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια χρονιά στην άλλη. Ε, σε ορισμένες χώρες μάλιστα τα πράγματα χειροτερεύουν. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Όταν θα συνεργαστείτε με τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα σας πρότεινα να προβλεφτεί κάποιο δεσμευτικό έγγραφο, ενδεχομένως κάποια οδηγία, κάποιο νομοθέτημα που θα αφορά στην μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διότι οι συστάσεις δεν αρκούν. Το βλέπουμε όλοι αυτό. Έχουν γίνει βεβαίως πολλά πράγματα θετικά, αλλά απευθύνομαι σε εσά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Ισταμπούλ ε, να ε, επικυρωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον 10 χώρε που δεν την έχουν επικυρώσει. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια προ την κατεύθυνση αυτή. Και τέλο, θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει υποστήριξη στο Ινστιτούτο για την Ισότητα των δύο φύλων, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, διότι αυτό το Ινστιτούτο είναι εξαιρετικά σημαντικό ε, για το σύνολο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Υπήρου είναι ένας θεσμός που πρέπει να έχει όμως και τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Όλοι αναμένουμε τη νέα στρατηγική και ελπίζουμε να μας παρουσιαστεί το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής μας ε, ε, η ομιλήτρια και τώρα η Εουχένια έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε που είστε εδώ κυρία Ιστόλα. Από ό,τι κατάλαβα στην ε, στρατική θέσμευση για το 2020 υπάρχουν τρεις γραμμές. Ε, η βία, η συμφιλίωση της, της και της ε, επαγγελματικής ζωής και η μισθολογική διαφορά. Χρειάζεται μια ομογενοποίηση της ε, νομοθεσίας, κάτι που δεν υπάρχει σε, ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν είναι και αποτελεσματική εφαρμογή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της βίας, έτσι, σε αυτό αναφέρομαι. Έγινε και σχετική αναφορά στην ανάγκη κυρώσεων και στην ανάγκη μιας μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας σε δικαστικό επίπεδο. Μας ανησυχεί επίσης ε, ότι ε, υπάρχει μια προσέγγιση ό,τι αφορά τη βία αυτή πολύ στενή και εδώ συμφωνώ με την ε, συνάδελφο σε ό,τι αφορά τη σύμβαση της Ισταμπούλ και την επικύρωσή της σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί μας απασχολεί ιδιαίτερα η σεξουαλική βία, όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις αμβλώσεις, ε, διότι η απαγόρευση της αμβλώσης είναι και αυτή η βία, είναι θεσμική βία. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη συμφιλίωση επαγγελματικής οικογενειακής ζωής, ξέρουμε, οπότε είπατε, δεν είναι αυτός ένας άξονα των εργασιών σας, ε, αλλά ποια είναι η άποψή σα για τις γονικές άδειε του πατέρα και της μητέρας και τη μητέρα που θα μπορούσαν ε, να προσμειώνονται 100% και οι δύο. Είναι στην πρώτη γραμμή στην Ισπανία αυτό ε, για κάποια πολιτικά κόμματα, είναι προτεραιότητα. Θεωρείτε ότι είναι εφικτή με τέτοια νομοθεσία. Μπορεί, αν δεν προχωρήσει με τέτοια νομοθεσία, πώς θα υπάρξει συμφιλίωση επαγγελματική και οικογενειακής ζωής. Ε, και σε ό,τι αφορά τις μυθολογικές αποκλήσεις ε, δίνεται μεγάλη έμφαση ε, στις γυναίκες, στα δυτικά συμβούλια, στα υψηλότερες ε, βαθμίδες, στις, Αλλά τι γίνεται με τις γυναίκες, παραδείγματος χάρη, που φροντίζουν ηλικιωμένους με πολύ πιο χαμηλούς μισθού. Αυτά, ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Γκάλβεθ Μουνιός έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για το έργο σας. Κυρία Ιστόλα, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Είπατε ε, ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες ε, και, και είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα. Ε, τα στατιστικά στοιχεία, και συγγνώμη που το τονίζω αυτό, ξέρω ότι τέθηκε ήδη, τα στατιστικά στοιχεία είναι εντελώ ανεπαρκή δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία για το Εράσμος, παραδείγματο χάρη, ή για άλλου τομεί. Ε, το βασικό πρόβλημα είναι, είναι ότι το στατιστικό μας σύστημα είναι γεμάτο στερεότυπα το ίδιο ε, και προωθεί τελικά τα στερεότυπα αυτά. Το ίδιο το στατιστικό σύστημα. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τη σωστή ανάλυση ούτε μια σωστή αξιολόγηση πολιτικής, της πολιτικής μας διότι δεν Έχουμε τα εργαλεία για να το κάνουμε αυτό. Θα ήθελα να ξέρω εάν υπάρχει πραγματική δέσμευση έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο θέμα της όρτας των δύο φίλων, διότι ακόμα και οι μελέτες, οι έρευνες που είναι σημαντικές για μια σειρά από θέματα όπως ε, η μισθολογική απόκληση, η στεξιωτική απόδειξη, απόκληση, ακόμα και η έρευνα αυτή βασίζεται σε ένα gentleman's agreement. Αυτό λέει η Eurostat για τις πληροφορίες που θα δίνουν οι επιχειρήσεις. Κάποιες χώρες ακολουθούν αυτές τις τάσεις κάποιες άλλες όχι, ε, καθυστερούν την ε, έρευνα αυτή ή, ή μειώνουν τόσο πολύ το δείγμα που δεν έχει νόημα. Είπατε ότι πρέπει να ηγηθούμε αυτών των στατιστικών στοιχείων για τα ε, για τις όνομες των δύο φύλων. Υπάρχει όμως ε, προϋπολογισμός για να γίνει κάτι τέτοιο. Σε επίπεδο κύριο Στάτ λέω, συγγνώμη που το ξαναρωτάω, υπάρχει πραγματική δέσμευση για να βελτιωθεί το στατιστικό σύστημα. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λίνα ο Ρόμπερτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Γενική Διευθύντρια που είναι εδώ μαζί μας σήμερα και για το έργο της. Τρία σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, η παρούσα κατάσταση ε, δεν βλέπουμε αλλαγές μετά τη σύμβαση ε, στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Ε, η βία, η ενδοκογενειακή, ε, τα σεξουαλικά δικαιώματα, δικαιώματα αναπαραγωγής, ε, τα δικαιώματα των LGBTI σε πολλές χώρες η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Έτσι για να το πω διπλωματικά. Και αναρωτιέμαι τελικά τι έχει συμβεί για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στα κράτη-μέλη. Και εσείς πώς, ως Γενική Διευθύντρια πώς ε, αντιλαμβάνεστε την κατάσταση αυτή όπου κάποια κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν καν στις συζητήσεις. Χρησιμοποιούν μάλιστα ε, πολύ σκληρά λόγια, ρητορική μίσους απέναντι σε κάποιες ομάδες. Ε, τώρα, για τα ίδια δικαιώματα στην αναπαραγωγή και τη σεξουαλικότητα, θα πρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα έχουν ίσα δικαιώματα, ίδια δικαιώματα στον τομέα αυτό και αυτό δεν συμβαίνει. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού και τι έχει γίνει για να εξασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση παραδείγματο χάρη σε νόμιμη άμβλωση ε, θα είναι νόμιμη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και όχι μόνο σε κάποια. Και βεβαίως ό,τι αφορά την οριζόντια ε, οδηγία κατά των διακρίσεων ξέρουμε ότι έχει μπλοκαριστεί εδώ και 10 χρόνια περίπου στο Συμβούλιο. Δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα και πρόκειται για μια σημαντική πρόταση έχει να κάνει με το mainstreaming σε όλους τους τομείς, όχι μόνο σε κάποιους. Όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι έχει γίνει για να εξασφαλίσουμε ότι η οδηγία, η οζόρια οδηγία κατά των διακρίσεων ε, θα εγκριθεί. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η Ελένη Φίτσον. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Γενική Διευθύντρια για την σαφή και εξαιρετική εισαγωγή τους. Θα ήθελα να τονίσω το ότι μιλάμε πολύ για την εξουσία, τη βία, τους μισθούς, αλλά η μεγάλη πρόκληση είναι ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι το 1 τρίτο των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εργάζεται γνωρίζουμε πως ε, όταν μια γυναίκα ε, μπορεί να δουλέψει ε, μπορεί να είναι ανεξάρτητη και αν σκεφτούμε πόσες γυναίκες δεν έχουν δικό τους εισόδημα θα ήθελα να είμαστε πιο σαφείς για την σχέση μεταξύ ισότητας και απασχόλησης γιατί το κλειδί στην ισότητα είναι η ατομική ελευθερία Έχω επίσης ένα ερώτημα για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε κάποιους παραγόντες. Μιλήσαμε για το μισθολογικό χάσμα που είναι πολύ μεγάλο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πολύ μικρότερο στη Σουηδία, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ε, ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι οι εξελίξεις που βλέπουμε στην Σουηδία, που μειώσαμε το μισθολογικό χάσμα, έχει συμβεί ουσιαστικά στο δημόσιο τομέα. Αυτό έγινε με πολιτικές αποφάσεις και λάβαμε την απόφαση ότι οποιοδήποτε ε, είναι δημόσιος υπάλληλο ε, θα πληρώνεται το ίδιο για την ίδια δουλειά και όλοι έχουν δικαίωμα σε πλήρη εργασία. Και οι γυναίκες εργάζονται με πλήρη απασχόληση και βεβαίως ε, Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Πώς ε, θα γίνει αυτή η σύνδεση με την στρατηγική της ισότητας για να έχουν και οι γυναίκες την δυνατότητα να έχουν δικαιό τους εισόδημα και να υπάρχει αυτός ο παράγοντας προώθησης του ζητήματος για να διδαχτούμε από τις βέλτιστες πρακτικές. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολλά θέματα. Μαρία Σοράγια Ράμος. Eh, Ευχαριστούμε, κυρία Γενική Διευθύντρια, που είστε εδώ. Έχω μια ερώτηση για την ε, βία, μάλλον για την ε, ισότητα μεταξύ των φίλων. Όταν ε, συγκεντρώνεται στοιχεία, ξέρετε ότι δεν υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων μεταξύ των 27 κρατών μελών. Τι δυσκολία έχετε λοιπόν όταν ε, συνδυάζετε τα γεγονότα, τα δεδομένα. Πώς συνδυάζετε τα στοιχεία για τα θύματα έμφυλης βίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ενδεχομένως να σχεδιάσουμε στρατηγικές για να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα. να δούμε κι εμείς ποια είναι τα πρώτα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και τώρα για την επιγραμμική βία. Ήθελα να μου πείτε, εάν η στρατηγική μπορεί να αντιμετωπίσει το πορνογραφικό υλικό που δωρεάν διατίθεται σε ανηλίκους. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρώτη επαφή που έχουν με την σεξουαλικότητα οι ανήλικοι τα παιδιά είναι μέσω αυτού του πορνογραφικού υλικού που προσφέρεται απλόχερα και πολλές φορές έχουν μια τελείως δεσταυλωμένη εικόνα για το τι είναι σεξουαλικότητα και η σεξουαλική επαφή. Βλέπουμε ότι οι δράστες σεξουαλικών ε, επιθέσεων γίνονται όλο ένα και νεότεροι. Κατεβαίνει ο μέσο όρο ηλικία. Πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό, έχει επιπτώσει και στην εφηλιβία. Ευχαριστούμε πολύ, ε, κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Γενική Διευθύντρια για την επίσκεψή σας. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη, γιατί μιλήσαμε για την πρόσβαση των γυναικών στα board, στα συμβούλια, ε, για την οδηγία του 2014 και την καταγραφή στοιχείων που είναι έξω οικονομικά. Υποχρεώνται ιδιωτικέ επιχειρήσεις να δώσουν στοιχεία για την θέση των γυναικών και την ε, εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια. Υπάρχει αξιολόγηση του πώ έχει υλοποιηθεί αυτή η οδηγία και αν όχι, Γενικώ, ξέρετε, αν αυξήθηκε ο αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Εμένα μου φαίνεται σοβαρό ε, ζήτημα για τι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Είναι ένα πάτημα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και χρειάζεται διαφάνεια στα δεδομένα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι τελείω διαφορετική και έχει να κάνει με την προστασία των γυναικών προσφύγων. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα. Έχουμε κανόνε για την προστασία των γυναικών προσφύγων και θα πρέπει να εφαρμόζονται. Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Πιτιέρνο. Και μετά θα θέσω και εγώ μια σύντομη ερώτηση. Και τέλος, με όλα αυτά τα ζητήματα, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Στόλα. Να προτείνω απλώς το εξή. Ξέρω ότι μπορείτε να απαντήσετε τέλεια και να καλύψετε όλα τα θέματα. Αλλά θα τη ζητήσω να μας απαντήσει και γραπτός, διότι έχουμε ε, αγγίξει τόσα διαφορετικά ζητήματα Τόσε πτυχέ που δεν είναι δυνατόν να τι καλύψουμε όλε. Είναι η πρώτη όμω συνεδρίαση τη Επιτροπή μα μετά το θερινέ διακοπέ. Είναι σαφέ ότι μα απασχολούν πάρα πολλά ζητήματα και πρέπει να εντείνουμε τι προσπαθίε μα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Γενική Διευθυντρία για την ε, προσέλευσή τη και τη δουλειά τη και την παρουσίαση που μα έκανε. Να σταθώ σύντομα σε μια ιδιαίτερη πτυχή της βία κατά των γυναικών βία σε δημοσίους χώρους. Διότι μεταξύ τεσσάρων τυχών έχουμε ένα πιο σημαντικό εργαλείο τελικά από τη δική μας νομοθεσία, της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολη. Τα προβλήματα σωστά τα έθεσαν οι συνάδελφοι. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει κύρωση τη Σύμβαση από όλε τι χώρε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη διάσταση της βίας σε δημόσιους χώρους, δημοσία και κυρίως στο επίπεδο του λόμπινγκ και των παρενοχλήσεων, εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι θοπία και ε, η παρενόχληση. Υπάρχουν διαφορές στην ομοθεσία των διαφόρων χωρών εδώ νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα εργαλείο δεσμευτικό, νομικό δεσμευτικό, όπως έγινε και με την ενδοοικογενειακή βία και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να υπάρξει ένα τέτοιο αυστηρό νομοθέτημα για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε και να αναχαιτήσουμε την βία, τη σεξουαλική παρενόχληση και την θοπία σε δημόσιου χώρου. Ξέρουμε τι σημασία έχουν πάρει οι δημόσιοι χώροι τα τελευταία χρόνια. Μιλάω για το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα τώρα, έτσι. Μιλάμε για ένα κόσμο εικονικό. Αλλάζει ακόμα και η ίδια η αντίληψη και η πραγματικότητα των δημοσίων χώρων. Χρειάζεται λοιπόν εδώ ένα εργαλείο στα ύψος των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τελείωσε ο κατάλογος, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, σας ε, δίνω ξανά τον λόγο, αγαπητοί συναδελφοί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι δεδομένα διαθέτει η Γενική Διεύθυνση δικαιοσύνη. για ανθρώπους με αναπηρίες που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Πρέπει να δούμε τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τα δικαιώματα των γυναικών πολλές φορές ε, υποβαθμίζονται. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα φύλλα και την ε, ισότητα των γυναικών και σε αυτό το τομέα. τι δεδομένα έχουμε για τον καταναγκασμό των γυναικών με αναπηρίες. I mentioned a network of gender equality. I'd be interested who is in and how uh, more or less uh, the whole composition takes place because those networks normally have a... Τα δίκτυα αυτά είναι ε, τα δίκτυα αυτά έχουν τα δικά του δεδομένα και θα ήταν καλό να μάθουμε λίγα περισσότερα για το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε το σχετικό δίκτυο που συλλέγει δεδομένα και μετά για τι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα τα θεσμικά όργανα, πρέπει εδώ να πετύχουμε πρόοδο. Το θέμα αυτό καθυστερεί. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για δύο νομοθετικές, ε, για δύο κοινοπληκτικέ θητείες. Ξέρω όλε τι προτάσει που πέρασαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να ξεμπλοκαριστεί το θέμα. Πρέπει να προχωρήσει. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα εδώ. Οπότε έχετε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων για τα ζητήματα όπου θα μπορούσε να υπάρξει γοργή πρόοδο εάν προχωρήσουμε. Και τώρα με όλες αυτές τις ερωτήσεις που σας φορτώσαμε σας δίνω το λόγο. Και σε αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής μας το είδατε. Πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε, πόσο θέλουμε να δώσουμε όθηση σε κάποια θέματα σε αυτή τη νέα κοινοβουλευτική θητεία. Σας παρακαλώ, κυρία Αστόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι επεξεργαζόμαστε μια στρατηγική. Έχουμε λοιπόν πολλά δεδομένα από την ε, δημόσια διαβούλευση, τη δουλειά που γίνεται εντός της ε, Κομισιόν με τους διαφόρους επιτρόπους και την συμβουλευτική μας ε, επιτροπή και τους ειδικού. Η δουλειά λοιπόν γίνεται. Ταυτόχρονα βεβαίως είναι αυτή η δουλειά και της μελλοντική επιτροπής και η επόμενη επιτροπή Λέω αυτό γιατί σε πολλά τα ερωτήματα που άκουσα το ερώτημα είναι τι κάνουμε στη στρατηγική, τι υπάρχει στρατηγική. Ε, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, αλλά φιλοδοξούμε να έχουμε μια ισχυρή στρατηγική. Και θα ήθελα να επανέλθω στο ότι παρά το ότι υπήρχε ε, μια στρατηγική ε, η οποία είχε κάποια επιτεύγματα. Ε, νομίζω ότι προσπαθούμε να πετύχουμε το θέμα αυτό, χάρη σε εσάς και τους συναδέλφους μου. Δεν καθόμαστε δηλαδή όλη μέρα στο γραφείο και δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, σε πολλά από τα ερωτήματα θα απαντήσω γραπτός. Λοιπόν, θα αναφερθώ τώρα στα υπόλοιπα. Ε, αν ε, ε, δείτε και τις σημειώσεις μου, θα καταλάβετε ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα, αλλά θα προσπαθήσω. λοιπόν, το τι κάνουμε συγκεκριμένα για τις γυναίκες στα ΔΣ. Είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη και τα τελευταία χρόνια είχαμε κάποιες καταστάσεις όπου εντάξει, θεωρήσαμε ότι το πράγμα δεν προχωράει. Τώρα με τη στήριξη της Γερμανίδας ε, Προέδρου ελπίζουμε να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Επίσης ε, θεωρώ ότι το θέμα αυτό αφορά και ε, τα, της πολιτικής. Τώρα για τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης ε, πολλά από αυτά τα ζητήματα θα ξέρετε ίσως πως ε, υπάρχει ένα ερώτημα από το Κοινοβούλιο προς το δικαστήριο για το τι θα γίνει στην περίπτωση όπου πολλά μέλη έχουν υπογράψει την σύμβαση και κάποια άλλα δεν την έχουν κυρώσει. Πώς ε, θα ψηφίσουν ε, στο Συμβούλιο για να μπορέσει να προχωρήσει και η Ένωση στην Σύμβαση. Είναι ένα νομικό ζήτημα λοιπόν που είναι ανοιχτό. Και φοβούμε ότι η απόφαση για προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έρθει αύριο μεθαύριο, αλλά θα συμβεί και μην ξεχνάμε ότι εφαρμόζεται σε πολλά οπότε πολλά από τα ερωτήματα που αφορούν την ε, παρενόχληση, την παρακολούθηση, την βία, από αυτά και τα περισσότερα έχουν κάποια σχετική νομοθεσία. Επίσης, ε, θεωρώ πως η σημερινή συζήτηση είναι συνεισφορά στην στρατηγική. Αυτά τα οποία είπατε σήμερα λοιπόν ε, θα τα λάβουμε υπόψη κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ε, και όλων των άλλων ε, ζητημάτων ε, και βεβαίως θα εισακουστούν οι επιθυμίες σας για το ΣΥΝΤΟ. Νομίζω ότι και αυτό ελπίζω να φανεί στην στρατηγική την οποία επεξεργαζόμαστε για την διαφάνεια των αμοιβών το τι θα γίνει μετά την διαφάνεια Ιδού η απορία Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει κάποια ισχυρή δεσμεύση για τα κορίτσια και πώς θα φαίνονται. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται βαρετό, αλλά είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Τώρα, για τις προδιαγραφές ε, και τη σχετική δουλειά. Όταν όλα τα μέρη έρχονται και συμφωνούν σε κάποιες προδιαγραφές, ε, προφανώς υπάρχει και η δέσμευση συνήθως. Αυτό είναι ευκολότερο στο εθνικό πόδι στο διεθνέ επίπεδο. Πρέπει να το δούμε, αλλά όπως είπα στην αρχή, δεν είναι τα πάντα θέμα νομοθεσία. και κάποια φορά πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Η κοινωνική εταίρη μετά και η εμπλοκή τους. Μα γίνεται ήδη αυτό. Συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων. Μία δύσκολη ερώτηση γιατί αφορά τα λεφτά. Αλλά πρέπει να πω τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες που καταρτίζονται ε, νομίζω ότι αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο και έχουμε τα μέσα να διαδώσουμε αυτές τις ε, πληροφορίες κυρώσεις. Η ποινική νομοθεσία είναι ένα πεδίο αρμοδιότητας ε, των κρατών μελών βασικά. Οπότε πρέπει να δούμε το πώς θα προχωρήσουμε και το τι είναι σωστό. Συμφωνώ προσωπικά ότι η βία σε οποιαδήποτε μορφή πρέπει να τιμωρείται και βεβαίως η βία κατά των γυναικών. Τώρα το πώς ε, θα γίνει αυτό σε διεθνές επίπεδο. Ε, η ισορροπία τώρα της ε, επαγγελματική με την προσωπική ζωή, γονική άδεια κτλ. Πρέπει να το δούμε τώρα αυτό. Πώς ε, θα εφαρμοστεί, πρέπει να δούμε προσεκτικά το πώς θα το κάνουν τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι αυτό σημαίνει τεράστια αλλαγή σε πολλές χώρες ε, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι άδεια που δεν μεταφέρεται και βεβαίω εγώ πάντα ζηλεύω τους Σουηδούς που το έχουν κάνει ε, ως Φιλανδέζα βεβαίως πάντα τους Σουηδούς ζηλεύουμε Αλλά αυτό δείχνει ότι είναι καλό και για τις επιχειρήσεις το να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες να εργάζονται. Η ηγεσία και το ότι δεν λαμβάνεται υπόψη είναι η δουλειά που γίνεται στο σπίτι. Νομίζω ακριβώς το θέμα της ισορροπίας, της δουλειάς και της ε, ζωής ήταν ακριβώς να δοθεί γυναίκες η δυνατότητα να μπουν στην αγορά εργασίας, να υπάρχει δηλαδή η επιλογή και να είναι και δυνατή οικονομικά, γιατί υπάρχει επιλογή σε πολλές περιπτώσεις, αλλά οικονομικά δεν γίνεται για πολλές οικογένειες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα που ακόμα είναι για να αποφασιστεί Τώρα, αν υπάρχει κάποια μεροληψία στα στατιστικά στοιχεία, εδώ πέρα έχουμε πάλι έναν τομέα που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενσωματώσουμε την πολιτική του φίλου. Αλλά η Eurostat είναι ένας τεράστιος μηχανισμός. Δηλαδή, αν ξέρετε το τι γίνεται ε, τα στατιστικά στοιχεία από όλε χώρες. Είναι και θέμα κόστους, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν λοιπόν αμέσω. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πολλές ερωτήσεις, πολλές. Για την αντίδραση, συμφωνώ, υπάρχει μία αντίδραση ε, και πρέπει να την αντιπαλέψουμε. Αναφέρατε και τα δικαιώματα ΛΟΑΔ, η Κομισιόν ε, παίζει πολύ ενεργό ρόλο και προσπαθεί να τα προωθήσει όλα αυτά. Παραγωγικά δικαιώματα. Είναι θέμα υγείας, ε, αλλά είναι και αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε εδώ πέρα είναι περιορισμένη η προσέγγιση μας. Ε, γενικά για τις διακρίσεις η οδηγία περί ισότητας Η Φιλανδική Προεδρία τώρα υποσχέθηκε να παίξει πολύ ενεργό ρόλο. Προσπαθούν να το προωθήσουν με το να έρθει η πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο. Ελπίζω λοιπόν να δοθεί μια νέα όθηση, αλλά ε, νομίζω πως η Κομισιόν είναι πολύ ε, δεσμευμένη εδώ πέρα για την νομοθεσία για τα εργασιακά και για το να έχει η γυναίκα μια δουλειά και όχι μόνο ένα δωμάτιο όπως έλεγε και η συγγραφέας ε, νομίζω είναι και αυτό ένα ζήτημα Λοιπόν, ε, για τις εταιρείε ε, και την οδηγία να αναφέρω κάτι και για την ποικιλομορφία γενικώ για τη σχετική χάρτα, αλλά ειδικά για τις γυναίκες. Υπάρχει η υποχρέωση να ενημερώνουν οι εταιρείε, αλλά ταυτόχρονα και σε διμερή Και μετά ε, υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί ένα θετικό κύκλο. Για τις ε, πρόσφυγες ε, γυναίκες, η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το κυνηγάει, υπάρχει κατάρτιση των ανθρώπων εκεί στις εγκαταστάσεις, στα στρατόπεδα. Α, κάνουμε πολλά, αλλά μάλλον όχι αρκετά. Η δημόσια παρενόχληση. Κοίταξε και εδώ πέρα Είναι κάτι που αφορά την εθνική νομοθεσία και είναι ευκολότερο να πούμε ότι υπάρχει κάποια τιμωρία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια δράση στο νομικό επίπεδο. Τώρα, για την αναπηρία και τις εκλογές, παραδείγματος χάρη σε ευρωεκλογές ε, που πέρασαν. Προσπάθησαμε να δούμε κάποια τέτοια ζητήματα και μετά αναφερθήκατε στο δίκτυο και στο ποιοι είναι ακριβώς. Είναι ειδικοί, δεν ξέρω ποιοι είναι ακριβώς τώρα. Αλλά θα επανέλθω και θα σας ενημερώσω. Αυτά και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσω γραπτός. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, ε, πολύ ζωηρή ε, ανταλλαγή απόψεων καλό είναι να μαθαίνουμε, με ένα του δεν, να μαθαίνουμε τι διακυβεύεται. Είμαι βέβαιη ότι θα είμαστε σε στενή επαφή κατά την προπαρασκευή ιδιαίτερα των ερωτήσεών μας, των ετοιμάτων μας προς ε, τους υπεύθυνους επιτρόπους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Κλείνει αυτό το σημείο της διάταξης, ε, το, διότι η επόμενη καλεσμένη μας περιμένει. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν έτσι ζωή. Η ανταλλαγή απόψεων ήταν όμως και απαραίτητη και πολύ καλή. Το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη είναι το σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων με την Καρλίν Σέλε. Είναι η υποψήφια ε, για διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας μεταξύ των δύο φύλων μετά την κυρία Λάγκμπακ ολοκληρώθηκε η θητεία της κυρίας Λάγκμπακ και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων ε, με την ε, διάδοχό της. και να μας πει τι ακριβώς ε, θα, θέλει, θα θέλεις να κάνεις στο μέλλον. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα σας δώσω το λόγο κυρία Σέλε για να κάνετε κάποια αγωγικά σχόλια. Συγγνώμη που περιμένατε έξω, αλλά βλέπετε εδώ έχουμε μια επιτροπή με μέλη τα οποία επιδεικνύουν εξαιρετική αυταπάρνηση και ε, ζήλο στα καθήκοντά τους. Γι' αυτό καθυστερούμε κιόλας λίγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι 50, ήταν 50 ετών και εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι ήταν περήφανη ε, που μπόρεσε να ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδέ. Ε, τη πήρε τέσσερα χρόνια για το διπλωμά τη και ήταν εκεί μεταξύ των συμφοιτητών τη που ήταν 23, 24 και αυτή ήταν 50. παντρεύτηκε όταν ήταν 18 σταμάτησε τη δουλειά της διότι αυτό ήταν η συνήθεια για μια παντρεμένη γυναίκα στη χώρα της είχε το πρώτο της παιδί στα 19 ο άντρας της ήταν αυτός ο οποίος εργαζόταν και αυτή ασχολούταν με την οικογένεια και τα οικιακά τα κατάφερε τελικά ναι πήρε το δίπλωμά της όταν ανακοίνωσε όμως την πρόθεσή της να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι το δίπλωμά της δεν θα της χρησιμεύσει κάτι. Δεν ήταν απαραίτητο για την οικογένειά της και αφού δεν ήταν απαραίτητο για την οικογένειά της, προφανώς δεν ήταν απαραίτητο και για αυτήν. Δεν σας έχω πει που συνέβη αυτό σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα συνέβη. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, σύμφωνα με τα δεδομένα του, το δείχνει αυτό. Τα στοιχεία για την αγορά εργασία δείχνουν ότι είναι 40% ο χρόνο εργασία τη γυναίκα σχέση με τον άντρα. Και υπάρχει μια 20, ένα 20% σε βάρο των γυναικών σε ό,τι αφορά τη μισθολογική απόκληση. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο τη ζωή των γυναικών και τι επιλογέ που κάνουν, αλλά και των οικογενειών τους τη ζωή. Οι δύο κόρες της ήταν εξαιρετικά περήφανες για τη, για τη μητέρα τους όταν πήρε το δίπλωμα, αποφάσισαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ήθελαν να είναι ανεξάρτητες, να έχουν το, τα δικά τους έσοδα και να βοηθήσουν άλλες γυναίκες, τις κόρες τους, τις συναδέλφους της, τις φίλες τους, για να κάνουν το ίδιο. αυτή η στιγμή, η στιγμή της αποφύτησης ε, ήταν το 1994 και η γυναίκα, η κόρη της μάλλον ξεκίνησε ως πολιτικό σύμβολο για κοινωνικά ζητήματα. Αυτή η γυναίκα για την οποία σας μιλάω είναι η μητέρα μου. Η δική της πραγματικότητα μου έδωσε κίνητρο να επιλέξω ε, το δικό μου δρόμο και στις σπουδέ μου και στη ζωή μου και με φέρνει εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, είναι τιμή μου ε, που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με καλέσατε από την ιδιότητά μου ως ε, υποψήφια για τη θέση της Διευθύντριας του Ινστιτούτου να σας πω ποιο είναι το δικό μου όραμα για αυτό που, μπορούμε να, αυτό που μπορεί να πετύχει το Ινστιτούτο στον τομέα της όρτας μεταξύ των δύο φίλων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Το πρώτο μήνυμά μου είναι το εξή. Πρέπει κάθε μέρα να υπάρχει ένας αντίκτυπος. Η κάθε μέρα, η εμπειρία της κάθε μέρας επηρεάζει τους ανθρώπους για τα ζητήματα αυτά. Το 2008 ως αναπληρώτρια ε, στη Γενική Διεύθυνση για την Ισότητα ε, και τα Δικαιώματα των ε, Ατόμων LGBT είχαμε σημειώσει σημαντική προδοτότητα στο Υπουργείο στο οποίο εργαζόμουν υπήρχε ένα σχέδιο υπήρχαν συγκεκριμένα μέσα και τα άλλα υπουργεία ήταν ικανοποιημένα με τις δράσεις μου, τις δράσεις μας. Όμως για μέρα του Οκτώβρη επισκέφθηκα ένα καταφύγιο για γυναίκες. Και τι είδα εκεί. Απελπισία. Οι γυναίκες αυτές είχαν χτυπηθεί από του άντρε τους, ορισμένε από αυτέ κάθε μέρα. Και ήταν εκεί στο καταφύγιο, σε ένα καθεστώς απόλυτης αβεβαιότητας, δεν είχαν πρόσβαση στα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, τα οποία τους είχαν αφαιρεθεί. Κάποιες άλλες δεν γνώριζαν που είναι τα παιδιά τους. Αν γύρισαν στις οικογένειές τους, ε, θα, είχαν, δεχόταν σαν πίεση για να επιτρέψουμε τους άντρες τους. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά από αυτό. Όλες αυτές οι ιστορίες, όλη αυτή η απελπισία με κυνηγούσε. Αυτή η επίσκεψη με οδήγησε στο ερώτημα πώς γίνεται ε, που όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη θέση μας δεν δείχνουν την πραγματικότητα αυτή. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς αυτές, ε, οι γυναίκες ε, μας είχαν διαφύγει από την πολιτική μας για την οποία ήμασταν τόσο περήφανοι. Πώς ήταν δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Πήγαμε σε άλλα υπουργεία, αρχίσαμε να κάνουμε μια αξιολόγηση των πολιτικών με βάση το φύλλο. Αν εφαρμόσουμε λοιπόν τις πολιτικές αυτές βήμα-βήμα σε άντρες και γυναίκες, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν πάρα πολλά κενά που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Αλλάξαμε κάποια πράγματα, μάθαμε. Είχαμε επικεντρωθεί μόνο στη μεγάλη εικόνα, όμως είναι και το ε, μέρους βήματα, οι συγκεκριμένες διαδικασίες, που και αυτές πρέπει να διέπονται από ένα όραμα που αφορά τα δύο φύλλα και την ισότητά τους. Είδαμε ότι υπήρχαν κενά σε αυτή τη μεγάλη εικόνα. Και έτσι αποφασίσαμε να λάβουμε δράση για να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο των πολιτικών μας. Το δεύτερο μήνυμά μου λοιπόν, σε ό,τι αφορά το όραμά μου, το τι μπορούμε να πετύχουμε δηλαδή, είναι ότι πρέπει να μπορούμε να κάνουμε zoom, να δούμε τι συμβαίνει ε, στην καθημερινότητα και να έχουμε και τη συνολική εικόνα. Έτσι μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε ε, τους, τους μας να βρουν τα κενά αυτά τους υπόλοιπους υπεύθυνου, πρέπει και να μπορούμε να μπούμε στη μικρή εικόνα ε, στις μεμονωμένες περιπτώσεις και στην μεγάλη εικόνα. Το 2012, μια μέρα χιονισμένη, υπήρχε μια επιτροπή του το των γυναικών ε, όπου συμμετείχαν και άτομα LGBT. Για πρώτη φορά περιμέναμε περίπου 30 άτομα. Ήρθε όμως ο διπλάσιος αριθμό, 60 άτομα. Ήταν προφανές ότι υπήρχαν κάποιε ομάδες ανθρώπων με διαφορετικέ απόψει για το θέμα αυτό. Και στην αρχή υπήρχε ένταση, υπήρχε σιωπή και αβεβαιότητα. Δύο πράγματα όμως άλλαξαν. Το πρώτο ήταν ότι παρουσιάσαμε δεδομένα, στοιχεία και τα στοιχεία έδειχναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε LGBT στην καθημερινότητά του. Και εκείνη τη μέρα κατάλαβα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά το πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα ανοίγουν το διάλογο. Οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι ε, έντονες, συγκινησιακές όμως και συναισθηματικές, αλλά τα δεδομένα μας επαναφέρουν στη λογική του διαλόγου. Κατέστησα φές εκείνη τη συνάντηση ότι πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις και επικράτησε ο σεβασμός δημιουργήθηκε εμπιστοσύνη και γαλήνη, ένας νέος άντρας σηκώθηκε και έκλαιγε. Μπόρεσε να μιλήσει για σεξουαλικό προσανατολισμό για πρώτη φορά στη ζωή του. Και το έκανε αυτό διότι αισθανόταν ασφαλής. Οι επικοδομητικές συζητήσεις αυτές εκείνης της μέρας με σημάδεψαν. Όλοι έχουμε απόψεις που είναι σημαντικές για μας είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ανταλλάσσουμε αυτές τις απόψεις, τις διαφορετικές απόψεις, να τις αντιπαραθέτουμε, σεβόμενοι όμως ο ένας τον άλλον. Και αυτή είναι η τρίτη ιδέα για το όρομά μου, για το τι μπορεί να κάνει το Ινστιτούτο για να πετύχουμε. Καθημερινός αντίκτυπος, αμοιβαίος σεβασμός, zoom στις μονομένες περιπτώσεις, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα όλοι μαζί. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ αυτά που είπε η, πρόεδρος, η νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στον τομέα της όρτας μεταξύ των δύο φύλων. Αναφέρθηκε σε, μια δίκαιη κατανομή για τις γυναίκες. Να δούμε λίγο τα στοιχεία. Τι μας δείχνουν τα στοιχεία για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στα κοινοβούλια. Το γράφημα δείχνει πόσες γυναίκες υπάρχουν στα κοινοβούλια της Ευρώπης τον 28 από 2004 βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόοδο, όπως βλέπει, όπως δείχνει η γαλάζια γραμμή, όμως εάν δεν αναλυφθεί κάποια δράση, η όταν δεν αναλαμβάνει τη δράση, μάλλον η πρόοδο είναι πιο αργή, κίτρινη γραμμή. Και όταν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές όπως οι ποσοστώσει, τότε η πρόοδο είναι πιο γρήγορη, πράσινη γραμμή. Με βάση τα δεδομένα αυτά και ακολουθώντα την μέση εξέλιξη, πότε θα έχουμε πλήρη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Πότε θα είναι πραγματικά δίκαιη η κατανομή. Σε 55 χρόνια πού θα είσαστε πιστεύετε το 2074. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το 2074 θα έχουμε φτάσει στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων εφόσον δεν αναλάβουμε καμία δράση. Και το 2048 πώς σας φαίνεται. Σε 20 χρόνια περίπου. Πόσο χρονών θα είναι οι κόρες σας, οι ανιψίες σας. Τόσο χρόνο θα μας πάρει για να φτάσουμε στην ισότητα των δύο φύλων. Ίση κατανομή λοιπόν με, τον, με τους παρόντες ρυθμού. Εάν αναλάβουμε δράση ακόμα και τώρα βλέπουμε ότι και πάλι πρέπει να περιμένουμε 16 χρόνια. Και μιλάμε τώρα για ποσοτικές πληροφορίες, έτσι. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η ποιοτική πτυχή του ζητήματος για τα κοινοβούλια. Αυτό είναι ένα τομέα. Ένα τομέα συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, μεταξύ πολλών στον τομέα τη των δύο φύλων. Ασχολούμαστε και με πολλά άλλα μέτρα πολλούς άλλους τομείς. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ανταλλάξουμε απόψεις από αυτόν σήμερα, ελπίζω. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να δείξουμε τα, επόμενα πέντε χρόνια ότι αναλάβαμε δράση για να κάνουμε τη διαφορά στον τομέα της ισότητας μεταξύ των δύο, των, των δύο φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, στο μέλλον να μπορούν να κοιτάξουν πίσω τους και να δουν τι πετύχαμε θα δουν, τι θα δουν τότε, θα δουν ε, άδεια καθίσματα ή θα έχει γίνει κάτι που θα έχει βελτιώσει τα πράγματα για το μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι το Ινστιτούτο μπορεί να φέρει παραδείγματα, δεδομένα, ιστορίες που θα βοηθήσουν για να έχουν πολιτικές που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο και την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. αυτό είναι το δικό μου όραμα για το Ινστιτούτο και το πώ το Ινστιτούτο μπορεί να υποστηρίξει το κοινοβούλιο αυτό τα επόμενα πέντε χρόνια για να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Όπω βλέπουμε, όπω δείτε στο γράφημα που μόλι σα έδειξα, χωρί εσά, χωρί εσάς, αυτό ο αντίκτυπο δεν είναι εφικτό. Περιμένω με ανυπομονησία να σας ακούσω, να καταλάβω ποιο είναι το δικό σας όραμα, οι δικές σας προσδοκίες. Εφόσον επιλεγώ, ε, αναμένω να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να κάνουμε τη διαφορά. Και φτάνω στο τελευταίο ερώτημα. Πώς μπορεί το Ινστιτούτο να σας βοηθήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας. Uh, thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την τόσο προσωπικά φορτισμένη παρουσίασή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο σε όλα τα μέλη που σήκωσαν το χέρι τους. Η κυρία Ραφαέλε, η πρώτη που ήθελε να θέσει ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά, αφού καλύπτονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και χαίρομαι ιδιαίτερος. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι τι θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει διαφορετικά το Ινστιτούτο υπό την δική σας ε, διεύθυνση σε σχέση με το παρελθόν. Και το δεύτερο είναι ότι με ενδιαφέρουν ε, πάρα πολύ τα θέματα διατομεακής ε, προσέγγισης ε, που αναπτύσσουμε καθώς συχνά είναι κάτι το οποίο λείπει. Να δούμε δηλαδή να αναγνωρίσουμε τις διαφορές μεταξύ γυναικών και να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Πώς θα φροντίσετε τα θέματα αυτά να αναδειχθούν περισσότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μελχιόρ. Ευχαριστώ που ήρθατε και για την τόσο παθιασμένη ομιλία σας μας ενέπνευσε. Υπάρχει πρόβλημα με τη βία κατά των γυναικών και πολλές φορές μιλάμε για σωματική βία που ε, συχνά είναι το, η δεύτερη συνέπεια της ψυχολογικής βίας. Εσείς Πώ το αντιμετωπίζετε αυτό στο επίπεδο του Ιδρύματο του Ινστιτούτου. Αναφέρατε την ανάγκη να έχουμε καλύτερα δεδομένα. Η δική μου εμπειρία από την προεκλογική μου εκστρατεία το 2014 ήταν ότι όταν το Ίδρυμα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εξέδωσε έκθεση για τη βία κατά των γυναικών, είδαμε ότι η Δανία έχει τεράστιο πρόβλημα με τη βία κατά των γυναικών. Κάτι που αντιφάσκει με τη δική μας την αντίληψη για την ίδια μας τη χώρα. Όμως δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα ακριβώς γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να ταυτιστεί με το αποτέλεσμα των ε, δεδομένων και της έκθεσης. Σε σχέση λοιπόν με το όσα ακούσαμε στην συζήτηση που προηγήθηκε. Πρέπει να συλλέγουμε δεδομένα με ακρίβεια για την ε, διάσταση των φύλων σε όλες τις πολιτικές. Πώς γίνεται να υποχρεώσουμε την Eurostat να κάνει το θέμα των γυναικών ε, πιο προβεβλημένο στη συλλογή δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ και τώρα θα κλείσω τον κατάλογο των εγωρτών. Η κυρία Περέιρα και η κυρία Σταράς Φεραγκούτ, η κυρία Άχο and uh, Maria Manuel uh, So με αυτές ε, τις παρεμβάσεις θα ολοκληρώσουμε. Κυρία Περέιρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Η ομάδα της ΓΚΟΕ ανέκαθεν συνεργαζόταν με το Ίδρυμά σας. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η σχέση τα επόμενα πέντε χρόνια. Κατά την άποψή μας είναι σημαντικό να καταπολεμήσουμε από κοινού την εμπορία ανθρώπων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την πορνογραφία, να προωθήσουμε τη σεξουαλική υγεία και τα αναπορικά δικαιώματα, καθώ και την ισότητα στο χώρο εργασία και την υγεία των ε, νεαρών γυναικών και κοριτσιών. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για τις πολιτικές απασχόλησης όπως εφαρμόζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και τη δημόσια δίκαια, διοίκηση χωρίς να λαμβάνουν υπόψη όμως τη διάσταση των φύλων και χωρί να κοιτάνε τι αντίκτυπο έχουν αρνητικό ή θετικό στον ε, αγορά εργασία. Έχουμε δείκτε για την μισθολογική ανισότητα στι δημόσιε υπηρεσίε και τη δημόσια διοίκηση. και τις δυνατότητες ανέλεξης, επαγγελματικής ε, ανέλεξης για άντρες και γυναίκες. Αυτοί οι δείκτες μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστούμε. Ρόζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Σέλε. Πολύ σύντομα είναι σημαντικό βέβαια στο θέμα των δύο φίλων σε όλη την Ένωση. Ε, η ισότητα δημιουργεί και ανάπτυξη, δημιουργεί ευκαιρίες για όλους, δημιουργεί μέλλον. Στο Ινστιτούτο λοιπόν που θα διευθύνεται ελπίζω σύντομα ε, προκύπτουν στατιστικά στοιχεία συγκριτικά μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ισότητα μεταξύ των φύλων. Είναι σημαντικό να έχουμε τα στοιχεία αυτά στη διάθεσή μα για να γνωρίζουμε επακριβώ πού λειτουργούν και πού δεν λειτουργούν τα πράγματα. Πού πρέπει να παρεύουμε και πού όχι. Και για να ανταλλάξουμε επίση βέλτιστε πρακτικέ. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα δημόσια χρήματα ε, που όταν διατίθενται λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των δύο φύλων και φτάνουν στου πολίτε ε, ισότιμα. Και αυτό βεβαίω επηρεάζει και τον προπολογισμό. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Το Ινστιτούτο είναι αυτό που μα παρέχει δεδομένα, αλλά δεν έχουμε αρκετά δεδομένα σε ό,τι αφορά τη συμφιλίωση ε, μεταξύ ε, και, οικο, και ζωής, ε, το sexting, ε, την, ε, τις νέες δυνατότητες, ε, προσεγγίσεις ό,τι αφορά την παρενόχληση, ε, το ψηφιακό χάσμα κτλ ε, λείπουν δεδομένα και για γυναίκες με ειδικές ανάγκες αναχώρα ε, και ποιες πρακτικές μπορούν να υπάρξουν. Κάτι με το οποίο συμφωνούμε όλοι, το θέμα της βίας ε, και τα δεδομένα για τη βία ε, ποιοι είναι οι τύποι βίας, ε, τι γίνεται με τον χρόνο ε, που έχουν οι γυναίκες αυτή τη στιγμή ε, την οποία καταγγέλουν, την οποία, και πώς μπορούμε να πετύχουμε τελικά αυτή την ισότητα, την ευκαιριών. Ευχαριστώ. Η Μαρία έχει τον λόγο. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ. Και χαίρομαι που παρουσιάζεστε και προσωπικά γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους, πρόσωπα που θα λαμβάνουν τις αποφάσεις και αν θα μπορούσα να σας ε, ψηφίσω θα σας ε, ψήφιζα. Κοιτάξτε τώρα, βλέπουμε το τι γίνεται στο Κοινοβούλιο από τα δεξιά με τις επιθέσεις, ε, με fake news, οπότε τα σοβαρά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και θα είναι πιο σημαντικά στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν ε, να συλλέγουμε δεδομένα τα οποία θα είναι πολύ αξιόπιστα και θα μπορούν να αντέχουν σε συζήτηση. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να σας πω πως η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν σας ε, ζηλεύω. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θα είχα μία προτεραιότητα. Η Ευρώπη είναι κατακαιρματισμένη όσον αφορά την νομοθεσία περί πορνείας. Έχουμε τη Γαλλία, έχουμε το σκανδιναβικό μοντέλο, στη Γερμανία έχουμε ένα πολύ φιλελεύθερο μοντέλο ε, που αφήνει πολλές πληγές. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν πολύ διαφορετικά δεδομένα. Να δούμε λοιπόν αφενός ποια θα είναι τα θετικά στοιχεία ενός σκανδιναβικού μοντέλου ή και αν έχει αρνητικά. Ε, στη Γερμανία έχουμε σκοτεινά θα έλεγα δεδομένα γιατί δεν είναι εύκολο να υπάρχει συλλογή στοιχείων, τι γίνεται στο πεζοδρόμιο, πώς στέλνονται από τον ένα οίκο ανοχή στον άλλο οι γυναίκες ε, εντό της Ευρώπης. Αυτό θα ήθελα να γνωρίζω προσωπικά και πολλές γυναίκες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί στο θέμα της πορνείας ε, μπορούμε να ε, κάνουμε κάτι μόνο αν έχουμε δεδομένα. Δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και σας ευχαριστώ για την δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστώ Ιρέν. Ευχαριστώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ και για την παρουσίασή σας επίσης που ήταν πραγματικά για όλους μας συγκλονιστική. Ε, τώρα, για το Ινστιτούτο. Προφανώς χρειαζόμαστε στοιχεία. Εγώ προσωπικά από το πρωί είναι κάτι για το οποίο δεν έχω ακούσει τίποτα. Είναι το θέμα της γύρανσης. Και εκεί υπάρχει μεγάλη ανισότητα. θα βρεθούν πολλές γυναίκες ε, μόνες τους, όλο και πιο μόνες, ε, ε, σε δύσκολη κατάσταση. Στο Ινστιτούτο λοιπόν υπάρχει κάτι που να προβλέπετε και που να παρακολουθεί, εν περιπτώσει, το θέμα της γύρανσης και το πώς αυτό επηρεάζει και σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών αυτή την πρόκληση την αντιμετωπίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και βεβαίως το άλλο είναι, δεν είναι οι γέροι, είναι οι νέοι. Ε, υπάρχει μια παρακολούθηση σε ό,τι αφορά τη βία των γυναικών ε, στο σχολικό ε, περιβάλλον έτσι ώστε από μικρή ηλικία να προλάβουμε να χτυπούν τα χώρια τα κορίτσια υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές και μια βάση δεδομένων που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Ρόμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από αυτά που είπε και η Μαρία, η οποία τώρα βγήκε, εάν μπορούσα και εγώ θα υπερψήφιζα. Αμέσως κιόλας. Μάλιστα, εργαστήκαμε επί του θέματος επί χρόνια μαζί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ξέρω πόσο θαραλέα και δυναμική είναι και ξέρω τη δική σας δουλειά από το Ινστιτούτο. Η παρουσίασή σας ήταν φανταστική, πάρα πολύ ωραία. Μια γρήγορη ερώτηση λοιπόν. Είναι πολλά τα κανθόδη ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και φαίνεται να μην βρίσκουμε λύση σε όλα τα κρατημέλη, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ε, πολιτική μας δράση. Έχουμε πολλές εμπειρίες. από αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων που ανέλαβαν και την Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Εγώ τουλάχιστον τα έχω ζήσει αυτά. Πώ μπορεί να γίνει περισσότερη δουλειά ε, σε επίπεδο επιμέρου χωρών. Και άλλη μια ερώτηση για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Τι μπορεί να κάνει το δικό σας Ινστιτούτο και να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι για να γίνει περισσότερη δουλειά στους άντρες. Οι άντρες έχουν πρόβλημα με τη βία. Συνήθως εκείνη είναι η πέτη και η αυτουργή της βίας κατά των γυναικών. Τι μπορεί να γίνει παραπάνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πάλι, μπράβο σας και είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα. Ευχαριστούμε η κυρία Μέντες. Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαιρετίζω την τόσο καλή σας και διεξοδική παρουσίαση. Μας δώσατε κάποιες πολύ καλές ιδέες για τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε και σωστά εντοπίσατε κάποια στοιχεία όπως οι ποσοστώσεις. Η εμπειρία μας έδειξε ότι μέσα σε μία διετία με ένα νόμο που εφαρμόσαμε μπορέσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στις δημόσιες υπηρεσίες. 23% στις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλη πρόοδος για το διάστημα 17 19. Για τις αμφιβολίες μου όμως, τους ενδιασμούς που ήθελα να σημειώσω εδώ σήμερα και να σας βοηθήσουν στο μελλοντικό σας έργο είναι πρώτον ε, ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την τεχνολογία. Οι γυναίκες είναι πάντοτε λιγότερες. Ε, μιλάμε για τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα ε, που φαίνεται να έχουν ένα καλό μέλλον βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αυτή την ανισότητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα όπως ήδη κάναμε σε άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και η δική μου, για να δώσουμε ε, κίνητρο στα νεαρά κορίτσια να πάνε προς αυτά τα επαγγέλματα, προς αυτή την επαγγελματική σταδιοδρομία. Και μια δεύτερη ερώτηση πολύ σύντομα και πάλι έχει να κάνει με τα δεδομένα, δεδομένα που εδώ αναφέρθηκαν επανειλημμένως από το πρωί, η δυνατότητα τα δεδομένα αυτά να μας επιτρέψουν να διακρίνουμε τη λεγόμενη πολλαπλή διακριτική μεταχείριση. Κάτι που δεν επιτρέπει να δούμε πόσο οι γυναίκες υποφέρουν απλώ επειδή είναι γυναίκες ή αν αυτό συνδέεται και με άλλε μορφέ διακριτικής μεταχείρισης ταυτόχρονα. Ε, αυτά είχα να σημειώσω. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσέλευσή σας και την παρουσίασή σας στη σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστούμε, Μαρία Μανουέλ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, οπότε είμαι πολύ γενναιόδορη αλλά πολύ σύντομα κυρία Κολτούρα. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Ε, συγχαρητήρια ε, για την παρουσίαση και ελπίζω να έχετε καλή θητεία αν και εφόσον επιλεγείτε. Δύο πολύ γρήγορες παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Το ένα πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν στα μέλη κράτη θεωρούμαστε ότι είμαστε πολιτισμένοι και προσπαθούμε για την ισότητα των φύλων, δεν δηλώνονται όλα τα περιστατικά. Τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Είτε από ταμπού, είτε από προβλήματα τα οποία βρίσκονται στα μέλη κράτη. Παραδείγματο χάρη είχαμε το πρόσφατο παράδειγμα που λέει 100 γυναίκες πέθαναν το 2019 στη Γαλλία και η υπουργό παίρνει τα μέτρα της. Είναι 100. Μήπως είναι 200 και δεν το ξέρουμε. Ε, και οι τραυματισμοί και όλα αυτά που δεν φτάνουν στο θάνατο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε να βοηθήσουμε τα μέλη κράτη έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να έχουμε τα πραγματικά στοιχεία στη βία. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, μήπως επειδή εμείς οι ενήλικες συζητάμε γενικώ για τα θέματα που αφορούν τη βία, την ενδοοικογενειακή βία, δεν είναι μόνο η γυναίκα, είναι και τα παιδιά που παρακολουθούν και που η βία συνεχίζεται. Είναι οι θύτε και τα θύματα και τα παιδιά παίρνουν το ρόλο. Μήπω θα έπρεπε να δούμε και το κομμάτι μέσα στην οικογένεια, πώς θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να εκπαιδευτούν είτε από τα σχολεία είτε προγράμματα έτσι ώστε να μην συνεχιστεί η βία. Και επειδή υπόθηκε και το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αφορά τα παιδιά, αφορά και τους ηλικιωμένους. Μήπως θα έπρεπε να το δούμε λίγο συνολικά και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα απαντήσω την πρώτη ερώτηση στα Ολλανδικά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας ε, λόγια και τις ερωτήσεις σας. Θα τις απαντήσω μία-μία και τις ερωτήσεις ε, που έχετε. Θα απαντήσω την πρώτη ερώτηση λοιπόν στα Ολλανδικά. Τι θα κάνει διαφορετικά το Ινστιτούτο. Θα τονίσω ότι σέβομαι πλήρως ε, την ομάδα, την διευθύντρια υπό την οποία ξεκίνησε το Ινστιτούτο και οικοδομήθηκε και το έκανε αυτό που είναι με τους ανθρώπους της. Και νομίζω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Βεβαίως, και αυτό ισχύει για κάθε οργανισμό, ε, πάντα μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις, ε, κάποια πράγματα να γίνουν διαφορετικά, αυτό ισχύει γενικώ. Και νομίζω πως ε, ένα από τα πράγματα τα οποία βλέπω στο Ινστιτούτο είναι ότι ε, υπάρχουν πληροφορίες πάρα πολλές οι οποίες δεν είναι αρκετά γνωστές. Δεν ξέρουμε τι θησαυρό δεδομένων έχουμε στο Ινστιτούτο αυτό. Λοιπόν, αν ε, πράγματι ε, με ορίσουν θα προσπαθήσω ακριβώς να τις ε, διαδώσω με έναν τρόπο που θα τις κάνει γνωστές. Λοιπόν, ένα από αυτά τα οποία παρατήρησα, γιατί έχω εργαστεί σε τέτοιους τομείς στο παρελθόν, είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτούν τα δεδομένα και να μεταφραστούν σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην εισαγωγή μου ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ε, να υπάρξει ένα αφήγημα, να αναφερόμαστε σε περιπτωσιολογία, να γίνει πιο ελκυστικό το θέμα δηλαδή και έτσι να μπορέσουμε να δούμε το τι υπάρχει πίσω από τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αριθμοί, ε, που μας δίνουν κάποιες πληροφορίες, αλλά υπάρχει μια ιστορία από πίσω τους. Ε. Λοιπόν, μιλάμε για αριθμούς, αλλά πίσω από τους αριθμούς αυτούς βρίσκονται άνθρωποι. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι αυτό το οποίο σκοπεύω να κάνω. Για την διατομιακή προσέγγιση, συμφωνώ μαζί σας ε, πλήρως, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, ε, όταν κάνουμε παραδείγματος χάρη μια ανάλυση για τη διάσταση των φύλων όταν ξεκινάει ένα έργο. Αν γίνεται κάτι σωστά το βλέπουμε γιατί βλέπουμε ότι ο μισός πληθυσμός είναι οι γυναίκες αλλά στην ομάδα γυναίκες και στην ομάδα άνδρες υπάρχουν ε, άνθρωποι με διάφορα χαρακτηριστικά και ε, ακριβώ για κάποιους από αυτούς είναι πιο δύσκολο να μπουν στην αγορά εργασίας. Αν δείτε λοιπόν στα δεδομένα μας βλέπουμε ότι οι γυναίκες με αναπηρία συμμετέχουν με 19%. 19% αυτών εργάζονται, ενώ οι άνδρες ανάπηροι είναι 28%. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να είσαι και γυναίκα και ανάπηρη ε, για να βρεις δουλειά. Και θεωρώ ότι το Ινστιτούτο αυτό μπορεί να βοηθήσει στη χάραξη πολιτικής όταν ακριβώς αναλύσει τα δεδομένα. Ξαναλέω, μιλάμε για 50% του πλαισμού, μια τεράστια ομάδα η οποία έχει τεράστια ποικιλομορφία. Οπότε για να σκίσουμε ε, σωστή πολιτική ε, είτε πρόκειται για ένα κράτος, είτε για μια ΜΚΟ, είτε για το κοινοβούλιο. Χρειάζεται ακριβώς αυτά τα δεδομένα. Και αυτή η διατομιακή προσέγγιση είναι ακριβώς ε, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η, η διεπιστημονική προσέγγιση, όπως είπατε επίσης, ε, η πολλαπλή διάκριση πράγματι υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και έχουμε ήδη ξεκινήσει, αν δείτε την σελίδα μας θα δείτε εκεί πέρα τα διάφορα δεδομένα που αφορούν στην, ε, την προσέγγιση. Παραδείγματος χάρη γίνεται ένας συνδυασμός μεταξύ ηλικίας ε, και θέσης στην αγορά εργασίας ή εισοδήματος και αν λοιπόν διοριστώ θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το πώς μπορούμε να το διευρύνουμε. Αυτό όπως είπα για να ε, συλλέγουμε τα δεδομένα για να μπορεί να ασκηθεί η καλύτερη πολιτική από τα κράτη-μέλη. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τα καλύτερα δυνατά δεδομένα. Μετά, οι ερωτήσεις για... Ναι, με συγχωρείτε, ε, θα μιλήσω τώρα αγγλικά. Είναι λίγο περίεργο να μιλάω και τα Ολλανδικά γιατί Σπανίω το κάνω, δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια εμπειρία. Λοιπόν, θα επανέλθω τώρα στα αγγλικά. Τα ζητήματα περί... και οι ερωτήσεις περί βίας. δεν θα το πρόβλημα. Η μία πραγματικότητα όταν συλλέγουμε δεδομένα για την βία είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικούς ε, ορισμούς ε, και συλλέγουμε διοικητικά δεδομένα από πολλές διαφορετικές ε, πηγές και καμιά φορά είναι δύσκολο να είναι συγκρίσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο και με το Ινστιτούτο το τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά από την άλλη αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα ότι συλλέγονται με διαφορετικό τρόπο τα δεδομένα στα κράτη-μέλη. Αν δεν ξέρω αν μπορώ να το αλλάξω. Ίσως κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις, λέγοντας το τι ε, χρειάζεται το Ινστιτούτο, ίσως ε, ε, επέλθει μια αλλαγή. Δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ σήμερα, αλλά ήταν κάτι το οποίο είχα δει όταν ήμουν στο ΔΣ του Ινστιτούτου και ξέρω ότι το Ινστιτούτο ε, βρίσκεται σε μια εσωτερική διαπάλεια. Δούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, η έκθεση της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πράγματι η Δανία ήταν στι ε, στις ε, τρεις κορυφές, το ίδιο και στην χώρα μου, στην Ολλανδία, όπου είδαμε ότι ε, ήμασταν ε, στην κορυφή μεταξύ των 28 κρατών μελών και σοκαριστήκαμε. Και μάλιστα η έρευνα αυτή έγινε μιλώντας στις γυναίκες. Ε, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό από το να συλλέγουμε διοικητικά δεδομένα. Ναι, πρέπει να τελειώνουμε, μάλιστα. Νομίζω ότι η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμένων ξεκαθάρισε ότι οι χώρε στην κορφή τη λίστα ήταν αυτέ οι οποίε τα, τα πάνε αρκετά καλά στην ισότητα των φύλων. Οπότε, μία από τι εξηγήσει ήταν ότι ε, ίσω οι γυναίκε νιώθουν ασφαλέστερε ε, στο να λένε αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, πρέπει να παραδεχτώ ότι σοκαριστήκαμε και στην Ολλανδία που ήμασταν στην κορφή τη λίστα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του να μιλάνε με γυναίκες. Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσω. τι μπορώ να πω άλλο. Για τον ρόλο των ανδρών. Νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά και αυτό θα ήθελα να πω ως γενική παρατήρηση για να κλείσω. Ένα από αυτά τα οποία διαπιστώνω είναι ότι εμένα πάντα μου προξενούσε έκπληξη το ότι ο κόσμος δεν βγαίνει ε, στο δρόμο λόγω της βίας που υπάρχει. Ότι δεν κατεβαίνουν ε, ε, σε απεργία για το μισθολογικό χάσμα. Θεωρώ ότι συμβαίνει γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει το τι συμβαίνει. Και όπως είπε και η Γενική Διευθύντρια, η ενημέρωση είναι ε, πάρα πολύ σημαντική. Ε, δεν μας αρέσει να μιλάμε για τον μισθό μας, γι' αυτό δεν κατεβαίνει ο κόσμος και σε διαδήλωση, γιατί δεν ξέρουν ότι βγάζουν λιγότερα τους άντρες. Οπότε η ενημέρωση είναι ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε μέσω της παροχής δεδομένων, του να λέμε ιστορίες, να πούμε δηλαδή το τι γίνεται στο θέμα της ισότητας. Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι πολλά σημαντικά θέματα στο τομέα της ισότητας. Αν διοριστώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να έχουμε ε, δεδομένα ουσιαστικά για να προωθήσουμε την ισότητα και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω γιατί είναι σαφές από τις ερωτήσεις σας πως το δέμα σας απασχολεί και πάλι σας είπα ότι αντιοριστώ αναμένω τη συνεργασία μαζί σα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. So, thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ για τα καθαρά σας λόγια, για την απαντήση στις ερωτήσεις μας. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε στο μέλλον στενά. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε την ανταλλαγή απόψεων λοιπόν και περάμε στο επόμενο σημείο τη μέσα διάταξη, το σημείο 6, Γενικό Προπολογισμό ε, για το έτος 2020. Ψηφίσαμε τις τροπολογίες το πρωί. Τώρα έχουμε την γνωμοδότηση που συνοδεύει το ψήφισμα. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην Φράνσες. Ευχαριστώ Πρόεδρε ως πρώην ε, ε, αναπληρώτρια πρωθυπουργό ε, αλλά και υπουργό δικαιοσύνη στην Ιρλανδία, θεωρώ ότι η δημοκρατία στην, στην Ευρώπη δεν είναι ολοκληρωμένη ό,τι αφορά την, τις γυναίκες, την αναγνώρισή τους, τη μεταχείρισή τους. Το είδαμε και σήμερα το πρωί και βεβαίως αναμένω να συνεργαστούμε ε, με υπομονησία ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε ε, χρήσιμες πρωτοβουλίες από αυτή την Επιτροπή. Όπως ξέρετε, η κυρία Ματέρα ήταν η συγκήτρια ε, για αυτή την έκθεση στην προηγούμενη θητεία. Ανέλαβα τώρα εγώ και ευχαριστώ να παρουσιάσω σήμερα ε, την γνωμοδότηση. Σήμερα ψηφίσαμε τις τροπολογίες του προπολογισμού το πρωί. Το σχέδιο ψηφίσματος όμως, το σχέδιο γνωμοδότησης μάλλον, ε, μας δίνει μια εικόνα για το τι αναμένουμε από τον επόμενο προπολογισμό από την προοπτική τη δικής μας Επιτροπής, τη Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Οι προτεραιότητε τις οποίες προωθούμε εμείς είναι πρώτα απ' όλα η ανεξάρτητη ε, διάθεση κονδυλίων για τα ζητήματα που μας απασχολούν, χρηματοδότηση ε, για δράσεις που έχουν να κάνουν με τη συνέχιση της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και της εμπορίας γυναικών είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στην Ευρώπη και την εφαρμογή βεβαίως της Ισταμπούλ. Ακούσαμε σήμερα για την βία, ακούσαμε πολλά ζητήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι. Ε, πρέπει να επικεντρωθούμε στη δημιουργία θέσεων απασχόληση και στην πρόσβαση στην αγορά εργασία για τις γυναίκες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Διότι γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στην εργασία. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγει κάποιος από τη φτώχεια και αυτό βεβαίως συνδυάζεται με μια σωστή φροντίδα των παιδιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες. Χρειάζονται λοιπόν χρήματα για να υποστηρίξουμε την οικονομική εξαρτησία των γυναικών αλλά και την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε για τι γυναίκε στον τομέα τη επιχειρηματικότητα και είναι σαφέ. Το έχουμε δει στην Ιρλανδία. Με τη σαφή υποστήριξη, με τη, με τη σωστή ε, υποστήριξη, σωστή κατάρτιση, ε, η διαφορά φαίνεται αμέσως. Ε, θα ήθελα ε, μέσω της νομοδότησης αυτής επίσης και της τροπολογίας του προπολογισμού να εξασφαλίσω ότι θα δοθεί έμφαση στη χρηματοδότηση για την ισότητα των δύο φύλων στην ψηφιακή οικονομία και στους τομείς των νέων τεχνολογιών. Ε, ένας νέος τομέας τεχνολογικός θα, θεωρητικά θα ήταν ένα φορέα ισότητα. Το αποτέλεσμα είναι όμω το αντίθετο. Είναι μειωμένη η συμμετοχή των γυναικών στι νέε τεχνολογίε, ιδιαίτερα στην κατάρτιση και στην απασχόληση. Μόλι 17% των ειδικών νέων τεχνολογιών είναι γυναίκε αυτή τη στιγμή και υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε για την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από 16 δισεκατομμύρια ε, έως και 16 δισεκατομμύρια εφόσον θα τι γυναίκες να, εισέλθουν σε αυτήν την ψηφιακή οικονομία. Είναι μια ένα θέμα τη εποχή μα και πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία προ την κατεύθυνση αυτή. Θέλω να είναι ισορροπημένη γνωμοδότηση, θέλω να καλύψω και τομεί όμω όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη χρηματοδότηση ε, για την ισότητα των δύο φύλων. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε ε, να εκμεταλλευόμαστε τι δυνατότητε των γυναικών και μπορούμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο εμεί στην Επιτροπή αυτή μέσω των αποφάσεών μα στο δημοσιονομικό τομέα. Είναι ατυχέ ότι ακόμα ε, δεν υπάρχει επαρκή οικονομική στήριξη και χρηματοδότηση για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και σχετικά ζητήματα, ε, θα πρέπει ε, επ' αυτού εμείς να επιμείνουμε. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει, έχει ασπαστεί την ιδέα ότι οι γυναίκες έχουν πολλά, πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουν στο με στην ισότητα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα που θα καλύπτει τις ανάγκες και των ανδρών και των γυναικών στην Επιτροπή αυτή πραγματικά σας ενθαρρύνω να βελτιώσετε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, να υποβάλλετε τροπολογίες πριν από τις 12 το μεσημέρι την Παρασκευή βέβαια. Αν θεωρείτε ότι κάτι λείπει, ότι είναι ελλειπές το κείμενο, στείλτε γνωμοδοτήσει και ε, τροπολογίες και με βέβαιο ότι θα τις ενσωματώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίσετε ότι δεν και πολύς χρόνος. Η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. <laughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ την συγκεκριά μας, την κυρία Φιτσέραλτ. και να υποστηρίξω το πολιτικό μήνυμα που πρόβαλε η συγκεντριά μας, θέλω να τονίσω το εξής. Ακριβώς η θέση των γυναικών στο χώρο των, ε, ε της τεχνολογίας της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Η θέση μας έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με τη δεκαετία του 90. Σε χώρες όπως η δική μου, την, ε, την ε, Πορτογαλία, οι γυναίκες έχουν σοβαρή θέση και πρόοδο ε, στο χώρο της επιστήμης, των πανεπιστημίων. Πρέπει να μπουν δυναμικά και στο χώρο των ICT. Οι περισσότερες δουλειές στο μέλλον όλες θα έλεγα, θα απαιτούν δεξιότητες ICT. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την τάση να μην πηγαίνουν προς τα και οι Ιδάλλως θα δημιουργήσουμε μια δομική ανισότητα, ε, πηγή ανισότητας για το μέλλον. Πρέπει να υπάρξει κατάλληλη κινητοποίηση στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε οι επικοινωνίες, η ηλεκτρονική, μηχανική, πληροφορική να διδάσκονται και στις εταιρείες να κοιτάνε να μην εγκαταλείπουν οι γυναίκε στα σταδιοδρομία του λόγω αποθάρρυνση και να πηγαίνουν σε άλλε δουλειέ. Οι μηχανικοί, όταν είναι γυναίκε, είναι πολύ καλά εκπαιδευμένε, αλλά κάποιε φορέ διακόπτουν την καριέρα του ή δεν ανελίσσονται, διότι στι τεχνολογικέ εταιρείε, για άλλου λόγου, στι μεγάλε εταιρείε tech, θα πάνε πολύ χειρότερα γυναίκες από τις άλλους τομείς. Έχουμε λοιπόν δύο ε, μέτωπα στα οποία πρέπει να πολεμήσουμε και στο χώρο της εκπαίδευσης και στο χώρο της απασχόλησης. Πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περισσότερα, περισσότερη δουλειά, περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και να έχουμε μια καλύτερη ισότητα των φίλων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που θέσατε αυτό το θέμα που μπορεί να μας αποσχολήσει και στην Επιτροπή μας στο μέλλον. Κάτι άλλο. Από ό,τι φαίνεται όχι. Φανταστική δουλειά. Θα συνεχίσουμε μαζί. Σε ευχαριστούμε Φράνσις. Α, με συγχωρείτε. Εγώ έχω κάτι να πω. Να ευχαριστήσω την συνάδελφο για την δουλειά στην εισηγησή τη. Συμφωνούμε μαζί τη ότι πρέπει να συνεχιστούν όλε οι δράσει που ασχολούνται με την αντιμετώπιση και την πρόληψη όλων των μορφών βία κατά των γυναικών, των παιδιών και των νέων. Αλλά για να υπάρξει σοβαρή καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, πρέπει μεταξύ άλλων μέτρων να προβλέψουμε ένα σύστημα συλλογή και ανάλυση δεδομένων συστηματικά, διαρκώ, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πηγές αυτής της μάστιγας και να ε, υπάρξει κατάλληλη πολιτική αντιμετώπισης αλλά και απαραίτητες κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές που θα προλάβουν τις πηγές της βίας ε, κατά των, των ε, νέων και των γυναικών. Πρέπει να υπάρξει και κατάλληλη οικονομική επικοδότηση για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες κοινωνικές, εργασιακές και μισθολογικές εντός των κατών μελών και η πηγή αυτή αυτής της ανισότητας πρέπει να χτυπηθεί στην ε, ε, ρίζα της, ε, διότι Αλλιώ το φαινόμενο αυτό δεν θα πάψει να υπάρχει. Πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη στους οργανισμούς που αναλύουν το φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό η δουλειά του Ευρωπαϊκού Στρατούτου για την Ισότητα των Φύλων και την καταπολέμηση τη διακριτική μεταχείριση έχει ένα καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει ένα εργότερο ρόλο στην ε, επιδίωξη των στόχων αυτών και για του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΙΑ, για την υγεία των ε, μητρών και των παιδιών. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω. Σας παρακαλώ, λίγο πιο αργά. να βελτιώσουν ας πούμε την υγεία των μητερών και των ε, παιδιών και εδώ πρέπει να ασχοληθούμε με την προστασία της υγείας και του μετρικού θυλασμού πράγματα που θα μπορούσαν εν μέρη να καλύψουν ε, τις ανησυχίες μας. Και για τις τροποποιήσεις που θέλουμε να υποβάλουμε, πρέπει κάτι να κάνουμε για την αντιμετώπιση ε, της ανισότητας και της διακριτική μεταχείρισης της βάρο των γυναικών. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν διαβάζουμε είναι λίγο θέμα εδώ να μιλάμε τόσο γρήγορα. Φράντσις, έχεις κάτι να προσθέσεις? Όχι, όχι. Νομίζω ότι ήταν σαφές ότι οι περισσότεροι στηρίζουν το ζουμί της έκθεσης. Ίσως λίγο τα θέματα του ICT να τα αναπτύξω παραπάνω, αλλά θα το συζητήσουμε τη συνάδελφο και το θέμα της πρόληψης. Ευχαρίστως να δώσουμε για μια ιδιαίτερη έμφαση στην ε, πρόληψη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους για τις συνεισφορές σας και με αυτά τα λίγα λόγια, όπως είπε στην παρουσίασή της, 4 Σεπτεμβρίου 2019, πολύ σύντομα, το μεσημέρι, Με συγχωρείτε 6 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, όχι σήμερα στις 12. Την Παρασκευή στις 12 λέγει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Προπολογισμού θα ψηφιστεί το θέμα στις 14 Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν ε, ανάγκη να ανασκουμποθούμε. Με αυτά τα λόγια έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της συνεδρίασής μας. Διάφορα, φτάσαμε στο σημείο των διαφόρων. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Ωραία. Ημερομηνία επόμενη συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση, 12 Σεπτεμβρίου, κοινή ε, συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ από τις 3.30 έως τις 6, πολύ σύντομη, και η επόμενη τακτική μας συνεδρίαση είναι στις 23 Σεπτεμβρίου. Από τις 3 έως τις 6.30 στις Βρυξέλλες και στις 24, δύο συνεχόμενες ημέρες, 24 Σεπτεμβρίου από τις 9 έως τις 12.30. Ελπίζω να σημειώσατε στις ατζέντες σας, τις ημερομηνίες. Και με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να κηρύξω την λήξη της σημερινής μας συνεδρίασης, πρώτης μετά την ε, θερινή διακοπή. Περνάμε στις συνεδρίαση των συντονιστών, κάποιους τους χρειαζόμαστε ακόμα για τους συντονιστές. Και παρακαλώ να φύγετε όλοι από την αίθουσα. Καλό σας απόγευμα, θα τα πούμε σύντομα. Οι συντονιστές να παραμείνουν μαζί με τους συνεργάτες τους. <clears throat> Θα περάσουμε αμέσως στη συνεδρίαση συντονιστών